<laughs> Allora, buonasera, se prendete posto cominciamo. Καθίστε για να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ, αν θέλετε. Το ordine del giorno è stato trasmesso per... Λοιπόν, για το σχέδιο μήνυσας διάταξης το λάβατε το σχέδιο διάταξης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ευχαριστώ του σταζιέρ που με τη γραμματεία ετοίμασαν το ενημερωτικό σημείωμα. Τώρα, αναφορικά με τα αυριανά για το διευθυντή της Όλαφ μας είπαν ότι οι πολιτικές ομάδες έχουν την πρόθεση να αναστείλουν αυτή την ψηφοφορία για την 9η Νοεμβρίου φέτος. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε παρακαλώ. Υπάρχει κάποιος από εσά ο οποίο θέλει να μιλήσει σχετικά. Όχι. Επιβεβαιώνεται λοιπόν. Πολύ καλά. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι γεγονό η αλλαγή τη ημερομηνία. Η ψηφοφορία θα γίνει συνεπώ στι 9 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Πολύ καλά. Α συνεχίσουμε. Φυσικά θα ενημερώσουμε σχετικά τους ψηφοφόρους ότι ανεβλήθη η ψηφοφορία για την 9 Νοεμβρίου, ώστε να μην περιμένουν άσκοπα. Με χαρά διαπιστώνω ότι έχετε την κάρτα σας για την ψηφοφορία. Στο σημείο 3 σημείες διάταξης θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τώρα, για τη διαδικασία επί των εγγύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε περίπτωση ε, προγραμμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Τόιτς. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και θα ήθελα από καρδιάς ιδιαίτερα τους ευρωβουλευτές των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών επίσης να ευχαριστήσω με που με υποστήριξαν στο έργο αυτό όταν συνέτασα αυτή τη γνωμοδότηση. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω για αυτή τη δουλειά τα μέλη της Επιτροπής. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην είναι σημαντικό. Ακόμα επιτραπέζει σε τίθενται μόνο σημαντικά θέματα. Μεταξύ αυτών όμως υπάρχουν πιο σημαντικά ζητήματα. Είναι λοιπόν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρει να συμμετάσχει σε αυτό το θέμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λάβει εντολή αντίστοιχα ώστε να μπορέσει να δράσει για την υποστήριξη προγραμμάτων και σχεδίων σε τρίτες χώρες. Η νέα γνωμοδότηση και οι τροπολογίες τροποποιούν την παλαιά πρόταση, την αρχική πρόταση. Τις περισσότερες τροπολογίες τις δέχτηκα και τις ενέταξα στην δική μου γνωμοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους συναδέφους τις τροπολογίες που τις υποστήριξαν να τις υπερψηφίσουν, να τις υποστηρίξουν και έτσι να βοηθήσουν με θετικό πνεύμα ώστε να βοηθηθεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο ρόλο της. Eh, Ευχαριστώ κύριε Ντόιτσο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία άμεσα. Αρχίζουμε λοιπόν με την τροπολογία υπαριθμών 1, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Δεν λειτουργεί το μηχανηματάκι μου. Δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Άλλαξα θέση και η θέση επίσης αυτή δεν λειτουργεί. Μπορείτε να υπολογίσετε ότι είμαι υπέρ, εν πάση Όλοι είναι υπέρ, κανένα κατά, δεν υπάρχουν και εποχέ. Ομόφωνα δεν έχω την κάρτα μου για να ψηφίσω. Την έχασα στο Στρασβούργο και δεν μπόρεσα να την αντικαταστήσω ακόμα. Αλλά θα σας πω τι ψηφίζω. Εντάξει. Πολύ καλά. Τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, άρχιτη πληροφορία ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, άρχιτη πληροφορία ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, άρχιτη ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. άρχιδη ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ε, πέρας ψηφοφορίας 21 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Συνεχίζουμε με την ημερησία διάταξη. Έχουμε τη συνέχεια με την άρνηση της απαλλαγής του 2008 της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Παρακαλώ, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ αν είναι δυνατόν, αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να έχουμε μια σύντομη ε, ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους. Διότι είδατε τη διαδρομή που ακολουθήσαμε στο επίπεδο της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Με συγχωρείτε. Δύο λεπτά, Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να μιλήσω αν μιλάτε γύρω. Λοιπόν, όπως σας είπα, υπήρξε πάγο σε ένα μέρος του προπολογισμού του Οργανισμού αστυνομία. Αυτό το παρακολουθήσαμε την τελευταία φορά όταν ψηφίστηκε ο προπολογισμό. Και τώρα τι, θα, τι κάνουμε τελικά. Είμαστε υπο, υποχρεωμένοι να κλείσουμε τους λογαριασμού ε, ε, πριν από το τέλος του χρόνου. Και ποιε θα είναι οι συνέπειε, ε, αυτού του κλεισίματος. Θα ήθελα να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να ακούσουμε τον Διευθυντή του Διοικητικού Συμβουλίου για να του κάνουμε ορισμένα ερωτήματα. Διότι ήρθε με τον νέο διεύθυνση του οργανισμού στις 12 Ιουλίου, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει και μας έστειλε ένα μήνυμα που το λάβατε όλοι φαντάζομαι, με τα γενικά στοιχεία που σας στείλαμε. Μετά την ακρόαση που έγινε του Διευθυντή, αλλά θα ήθελα η Επιτροπή μας να υποβάλει ορισμένα ερωτήματα. Ήδη η Επιτροπή, το Δικό Συμβούλιο ε, έλαβε τα ε, ζητήματα την ΟΛΑΦ. Εμεί όμω δεν λάβαμε τα πορίσματα αυτής της έρευνας. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Λοιπόν, θα θέλαμε τουλάχιστον να γνωρίζουμε ποια ήταν τα πορίσματα της έρευνας. Ζητήσαμε ορισμένα ορισμένε πληροφορίε σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διαφάνεια για τα μέλη που απαρτίζουν αυτό το Συμβούλιο. Δεν μας το δώσανε. Μας είπαν ότι δεν μπορούμε να ε, αναρτήσουμε στο διαδίκτυο τα άτομα και ρωτώ γιατί. Γιατί δεν θέλουν τα άτομα αυτά να βλέπουν το όνομά του στο διαδίκτυο, ενώ σε άλλου οργανισμού τα ονόματα ε, των μελών του Διοικητού Συμβουλίου δημοσιοποιούνται. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εξαίρεση στον κανόνα και τι έγινε. Τι έγινε σε διοικητικό επίπεδο, ε, τι, απέναντι στον παλιό διευθυντή. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που θέλουμε να υποβάλουμε στον παλιό διευθυντή. Γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσω μαζί σα και να δούμε τι πιστεύετε κι εσεί. Δεν βιαζόμαστε, έχουμε ακόμα δύο μήνε. Μπορούμε να τον ακούσουμε τον Νοέμβριο, ή τον Δεκέμβριο και να προτείνουμε να κλείσουν λογαριασμοί πριν από το τέλο του χρόνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάζη το λόγο. πρέπει να πω ότι αυτό που είπε η κυρία Μάτιο είχαμε πολύ καλά συνεργαστεί ούτως ή άλλως και στη δουλειά για την έκθεση αυτή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία εκκρεμούν. Τα αναφέρατε αυτά κυρία Μάτιο και θα ήθελα να παρακαλέσω σχετικά τα άτομα αυτά να μπορέσουμε να τα συναντήσουμε ώστε να γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ κυρία Ματιό. Είστε d'accordo con, con la Prego. Ε, Πρόεδρε, δεν έχω καμιά αντίρρηση γι' αυτό. Πρέπει σίγουρα με αυτή την περίπτωση της ΕΠΟΛ να δώσουμε κάποια συνέχεια και να ασχοληθούμε παραπέρα. Πήρα την ελευθερία ως Ευρωβουλευτής ε, το θέμα αυτό να το απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κοινοβουλευτική ερώτηση. Τι σκέπτεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και οι συνθήκες απλά δεν προβλέπουν τίποτα για την περίπτωση αυτή για έναν οργανισμό, για μια υπηρεσία που αρνούμαστε εμείς να τις χορηγήσουμε απαλλαγή. Τι γίνεται τότε. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα πρόβλημα. Το αφήνει ανοιχτό και εκκρεμεί από πλευρά της συνθήκης. Είναι ένα κενό θα έλεγα. Ένα χάσμα. Θα χαιρόμουν αν θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Καμιά φορά οι απαντήσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όπως οι χρησμοί του μαντίου των Δελφών. Πρέπει να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Με ενδιαφέρει το θέμα της συνέχειας του ΣΕΠΟΛ που θα μπορούσε να τύχει συνέχεια από πλευράς επόμενου εισηγητή. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ή είναι εντάξει έτσι τα πράγματα. Ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, είναι το σημείο 5. Δεν ξέρω τι αποφασίσαμε, αλλά υπήρξε αυτό το αίτημα της κυρίας Ματιέ. Α, ωραία, ωραία, αναβάλλεται. Εντάξει. Εντάξει, ας κάνουμε μια προσπάθεια να συναντηθούμε με Διευθυντή. Εντάξει λοιπόν το θεωρούσα δεδομένο. Το άλλο σημείο στην ημερησία διάταξη Σήμερα έχουμε την ε, αναχώρηση αντιπροσωπεία στην Ιταλία. Θα γίνει η τρίτη συνάντηση τη αντιπροσωπεία μετά από τι σημαντικέ επισκέψει που έγιναν στην Ελλάδα και στην Κροατία. Πιστεύω ότι όλοι σα έχετε το πρόγραμμα που δεν είναι ακόμα οριστικό γιατί δεν μας έχει δοθεί η επιβεβαίωση της παρουσίας του, του, του Υπουργού Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας ε, Τρεμόντι ο οποίος επιφυλάχθηκε να διορίσει κάποιον που θα τον αντικαταστήσει, να ορίσει κάποιον που θα τον αντικαταστήσει. Το έχετε νομίζω το πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, μήπως κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Διαφορετικά συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμησης της απάτης, της γνωστής Όλαφ. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας... Παρακαλώ, κύριο Γκέι. Συγγνώμη πρόεδρε, ίσως πήγατε υπερβολικά γρήγορα ή εγώ είμαι υπερβολικά βραδύς, αργός σήμερα, δεν το ξέρω. Πολύ σύντομα θα ήθελα μια και δεν πιέζει τόσο πολύ τεράστια ο χρόνος να μιλήσουμε για την αποστολή αυτή της αντιπροσωπείας μας. Κάπως ανησυχώ πρόεδρε. Ανησυχώ για το τηλεοπτικό συνεργείο που μας ε, συνοδεύει στις εργασίες μας. Θα ήθελα να βεβαιωθώ σε αυτόν τον κύκλο από πλευρά σας αν έχει αποσαφινιστεί πού και σε ποια τμήματα του προγράμματος μπορεί να συμμετάσχει αυτό το τηλεοπτικό συνεργείο και σε ποια τμήματα όχι στη συνάντηση των συντονιστών ε, σε σχέση με, εξωτερι... Ε, σε σχέση με εξωτερικές ε, τέτοιες, τέτοια γυρίσματα νομίζω δεν τίθεται ε, πρόβλημα και το γραφείο ερευνητικών δραστηριοτήτων δημοσιογραφικών που ε, μπορεί να έχει επαφή με τις αντιπροσωπείες εφόσον υπάρχει προθυμία από πλευρά τους ήταν όμως σαφές σε εσωτερικές συζητήσεις ότι δεν θα συμμετέχει στις εσωτερικές μας συζητήσεις. Συμβαίνει αυτό ή όχι. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι τα πράγματα. Ήδη την προηγούμενη φορά αποφασίσαμε ότι ο τύπος δεν θα πάρει μέρος στις εσωτερικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Όπως το θυμούνται οι συνάδελφοι, γράψαμε μία επιστολή στους Βρετανούς δημοσιογράφους που ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνάντηση. Δεν μας ε, δόθηκε μία απάντηση, αλλά ε, ε, να επαναλάβω ότι ο τύπος δεν μπορεί να πάρει μέρος στις θεσμικές εργασίες της Επιτροπής. Ο τύπος θα, παρουσιαστεί στο, θα περιοριστεί στο να τραβήξουν ε, κάτι πριν από την ε, συνάντηση. Νομίζω ότι αυτή ήταν η συμφωνία μας. Ο κύριος Γκρές. Σας ευχαριστώ διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Πρέπει ο εμπιστευτικό χαρακτήρα ε, των διαβουλεύσεων μα να διασφαλιστεί. Εγώ χαίρομαι για το ιδρυτικό μέλο τη Ιταλία που θα πάμε εκεί αποστολή. Χαίρομαι για αυτή την αποστολή. Μπορούμε κάποια θέματα με το Υπουργείο Οικονομικών να τα συζητήσουμε, κάποια προβλήματα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Αν δεν κάνω λάθο, στου συντονιστέ και μια ακρόαση των υποψηφίων για την Όλαφ και κλεισμένων των θυρών την είχαμε συμφωνήσει δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι και το οποίο μου διέφυγε ή αν υπάρχει κάτι για το οποίο δεν θυμάμαι αρκετά καλά. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Είπαμε ότι και το hearing έτσι θα γίνει, αλλά είναι ήδη αργά τώρα πλέον. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε ένα πράγμα μόνο για για την προπαρασκευή, το υλικό για την προπαρασκευή. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού που σήμερα μας δόθηκε ακριβώς για την αποστολή στην Ιταλία είναι στα Ιταλικά μόνο. Και με κάθε σεβασμό για τον Ιταλικό λαό και την Ιταλική γλώσσα δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει κανείς Ιταλικά για να, να εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ξέρω ποιο είναι το καθεστώς αυτού του υλικού. Πώς διατέθηκε έτσι. Διότι αν συμπεριλαμβάνεται κάτι για το οποίο αναμένεται ότι εμείς θα πρέπει να το γνωρίζουμε, ε, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Αν είναι κάποιε λεπτομέρειε που δεν είναι υποχρεωτικό να τι γνωρίζουμε, εντάξει, τότε να δεχτούμε ότι μπορεί και να τι αγνοούμε. Η κυρία Καστίγιο, όπως ε, εσείς έτσι και εγώ είχαμε στα χέρια μας αυτό το υλικό που έφτασε καθυστερημένα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει κάποια μετάφραση. Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο. Θα έπρεπε το υλικό αυτό να το έχουμε έγκαιρα στη διάθεσή μας και με λυπή που δεν το είχαμε. Άλλες παρεμβάσεις για την επίσκεψη στην Ιταλία. Όχι. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ακρόασης των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Όλαφ. Όπως γνωρίζετε, έχουμε έξι υποψήφιους, τους οποίους θα πρέπει να ακούσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Όπως αποφασίσαμε σήμερα, παραπέμπεται η ψηφοφορία για τις 9 Νοεμβρίου. Αυτό που είναι σημαντικό για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στις ε, ακροάσεις αλλά και για να κριθούν υποψήφοι πάνω στην ίδια βάση ο κάθε ένας από μας θα πρέπει να σέβεται τους προβλεπόμενους χρόνους. Πέντε λεπτά για κάθε υποψήφιο. Έχει στη διαθεσή του λοιπόν πέντε λεπτά για να πει ό,τι έχει να πει μετά το πέρας των 5 λεπτών θα του αφαιρέσουμε το λόγο και μετά θα διατυπωθούν ερωτήσεις από τους διάφορους συναδέλφους. Τα ονόματά τους ήδη τα έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε ένα λεπτό για την απάντηση και προβλέπονται δύο λεπτά, για την ερώτηση με και προβλέπονται δύο λεπτά για την απάντηση. Η μέθοδος του πινκ-πονγκ. Ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση. Έχουμε ανάμεσά μας τον πρώτο υποψήφιο, ο κύριος Έρμπερτ Μπόσο που θα ήθελα να χαιρετήσω. Ο κύριος Μπόσο είναι δίπλα μου και μπορεί να μας κάνει άμεσα την παρουσίασή του. Να του θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι έχει πέντε λεπτά καιρό στη διάθεσή του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερο προνόμιο για άλλη μια ακομα φορα οτι εχει πεντε λεπτα καιρο στη διαθεση του ευχαριστω σα ευχαριστω πολυ προεδρε ειναι ιδιαιτερο προνομιο για αλλη μια φορα να κάθομαι σε αυτό το κάθισμα και ίσως πιο νευρικός από ό,τι στο παρελθόν, αλλά είναι πολύ πιο ευχάριστη αυτή η εμπειρία. Γιατί είμαι υποψήφιος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτον, ο, ο θλιβερός λόγος ότι ο πρώην Γενικός Διευθυντής ε, απεβίωσε υπερβολικά πρόημα. Δεύτερον, το ότι αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε τη μεταρρύθμιση της Όλαφ που πρόκειται να γίνει. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί κάθε μέρα να αναθεωρείται και να μεταρρυθμίζεται η Όλαφ. Γι' αυτό είναι ένα ιστορικό σημείο, ένα θέμα που με τον νέο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να ευθυγραμμιστεί και με τη μεταρρύθμιση. Και τρίτον, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να μπορεί κανείς με διάφορες ακροάσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αυτή την εμπειρία με τις ε, ημερήσιες αξιολογήσεις ε, χαρτοφυλακίων, υποψηφίων και έτσι χαίρομαι που είμαι εδώ υποψήφιος ενώπιόν σας. Τώρα, αν όπως γνωρίζετε ίσως ήμουν αρμόδιος εισηγητής σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο όταν είχαμε την εξέταση κάποιων ε, παρατυπιών ως περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε, de facto, είμαστε μια εξεταστική επιτροπή που λειτουργήσαμε επί αρκετούς μήνες και θα έλεγα υπό το δικό μου πρίσμα ήταν η πιο σημαντική μου διακριβωτική έρευνα αυτή. Τότε ως εισηγητής είχα και την ευκαιρία τους μηχανισμούς για την καταπολέμηση απατών και ατασταλιών να τους ε, εξετάσω σε βάθος και δεν ξεκινήσαμε από μηδενικό σημείο, κάτι υπήρχε ήδη προηγούμενα. Αλλά παρέμεινε παράλληλα με την Όλαφ το ότι από αυτή, τη, από αυτή την περίοδο που εμείς ως Κοινοβούλιο ε, είχαμε παρακολουθήσει τις δραστηριότητες, δύο σημεία είναι σημαντικά. Πρώτον, είναι επικίνδυνο στον τομέα της καταπολέμησης απατών όταν ε, δημιουργεί κανείς προσδοκίες που δεν μπορεί να τις ε, τηρήσει και στη συνέχεια τις αθετεί όταν δεν έχει τις σωστές αρμοδιότητες και δεν έχει την δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες. Τότε είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν οι προσδοκίες αυτές. Και αυτό πλήττει και το κίνητρο που έχουν οι συνεργάτες για να εργαστούν αποτελεσματικά. Και έτσι πρέπει να λάβουμε υπόψη και συμβιβασμούς ε, που πρέπει να ε, συνάπτονται. Δεύτερον, το θέμα της ευθύνης ή της υπευθυνότητας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό η προσωπική ευθύνη να την επομίζονται τα άτομα. Και στο τέλος, αυτό ήταν ένας από τους κύριους λόγους της κρίσης τη δεκαετία του 90 που δεν μου αρέσει υποχρεωτικά και οπωσδήποτε ο σημερινός μηχανισμός της Όλαφ που πολλά πράγματα ισοπεδωτικά τα αντιμετωπίζει. Πάντα μάθαμε μαθαίνουμε ότι στο τέλος κανένας δεν επομίζεται τις ευθύνες ή όταν πολλοί θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι τότε δεν υπάρχει κάποια ευθύνη που να μπορεί κανείς να προσωποποιήσει ε, υπεκφεύγει λοιπόν η ευθύνη και για την νομική πτυχή για το νομικό πρίσμα είναι τόσο πιο σημαντικό ακόμα το manpower τα στελέχη που εργάζονται στην Όλαφ να, μπορούν να, τα χρησιμοποιήσει, να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά μπορώ να σας διασφαλίσω ότι κάθε περίπτωση από τους επαΐοντες ε, θα εξετάζεται σε βάθος ε, για να φωτιστεί. Τώρα θα περάσω σε μια άλλη γλώσσα για να σας μιλήσω. Σας υπέβαλα προηγούμενα στο παρελθόν ένα σύντομο έγγραφο με τις απόψεις μου, τις ιδέες μου όσον αφορά την Όλαφ. Όπως προανέφερα, μάλιστα, ναι, η κυριότερη προτεραιότητα πιστεύω εγώ για τον νέο διευθυντή είναι η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της Όλαφ και βλέπω τον εαυτό μου και την υποψηφιότητά μου ως ένα υποψήφιο σε ένα άτομο που θα λειτουργήσει και θα δράσει για τη μεταρρύθμιση της Όλαφ. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το κυριότερο, το πιο σημαντικό σημείο. Έχουμε μια νέα συνθήκη που μας δίνει αρμοδιότητες, πολλές ευκαιρίες που δεν είχαμε στο παρελθόν για να δράσουμε και με το αντίστοιχο άρθρο της συνθήκης Λισαβόνας που είναι πολύ καλύτερο από εκείνο το οποίο είχαμε στο παρελθόν μπορούμε να δράσουμε σωστά. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί λοιπόν εσωτερικά, αποτελεσματικά η Όλαφ για να μπορεί να επικεντρώνεται στις έρευνες. Είναι ένα λάθος το ότι ένα τρίτο των στελεχών εργάζεται στον ερευνητικό τομέα. Ο δικός μου στόχος θα είναι για μια πενταετία τουλάχιστον 50% του προσωπικού της Όλαφ να ερευνά περιπτώσεις δραστήρια. Και ένα τρίτο σημείο. Πρέπει να αναθεωρήσουμε, να ξαναδούμε το νέο πλαίσιο τη νέα δουλειά και συνεργασία μεταξύ Όλαφ και του εισαγγελέα του δημοσίου κατηγόρου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε σε σχέση με τη συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Μπόσισο για την ομιλία σας. Ξεκινάει τώρα ο κύκλος με τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τη συνάδελφο Γκρέσ. Ένα λεπτό. Μάλιστα, σας ευχαριστώ και έτσι περνάμε ωραία και με ένα νέο ρόλο που είναι δυνατόν να αναλυθεί. Είδαμε τις κύριες αδυναμίες ε, όσον αφορά την υπηρεσία και τις ε, ερευνητικές δραστηριότητες και την παραγραφή λόγω μεγάλου διαστήματος που περνά. Και γι' αυτό στην προκήρυξη θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να επιλέξουμε ένα άτομο που έχει σε βάθος γνώση στον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι ευχάριστη τώρα έκπληξη αγαπητέ συνάδελφε να σας βλέπουμε ως υποψήφιο εδώ ενώπιόν μας και ίσως θα μπορούσε αυτό να εξηγηθεί πώς σε σχέση με το κείμενο της προκήρυξης εσείς ευθυγραμμίζεστε ως υποψήφιος σε σχέση με την προκήρυξή μας. Σας ευχαριστώ. Uh, να απαντήσω. Well, I think it's up to you to... Νομίζω ότι εναπόκειται σε εσά να το διευκρινίσετε αυτό με την Επιτροπή. Γιατί ο κατάλογος των υποψηφιωτήτων υπευλήθη από την Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων και πάλι. Είναι θέμα των θεσμικών οργάνων αυτό. Τα θεσμικά όργανα θα αποφασίσουν. Εγώ υπέβαλα την άποψή μου στα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Είμαι έμπειρος στην καταπολέμηση της απάτης, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, και θα είμαι υποψήφιος και τέρος για τα θεσμικά όργανα για να μπορέσει να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση. Μπορεί να είναι βοηθός, εταίρος. Η μεταρρύθμιση θα γίνει από τα όργανα. Γκέιρ. Αγαπητέ Χέμπερτ, καλώς ήρθες και από πλευράς μου σε αυτό τον κύκλο εδώ, στην Επιτροπή μας. Όταν πρόκειται για την όλα τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο με ιδιαίτερο βάρος και αξία στο θεσμικό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το συσχετισμό των θεσμικών οργάνων, των παλαιών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Μπορείς να μας εξηγήσεις από πλευρά σου πώς η πείρα σου στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεισφέρει όσον αφορά τη συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ θα ήθελα να μου επαναλάβεις τι, τι εννοείς. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η πείρα που έχεις σε σχέση με την συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα που για τον διευθυντή, τον γενικό διευθυντή του Όλαφ αυτό θα αποτελούσε ιδιαίτερη πρόκληση. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Γνωρίζετε ότι δεν το ανέφερα πιο πριν, αλλά η Όλαφ βασίζεται σε σχέση με μια έκθεση που εγώ είχα συντάξει στο παρελθόν ως αρμόδιος εισηγητής για αυτές τις δραστηριότητες και στις διαπραγματεύσεις υπήρξε αναζωογόνηση σε καθημερινή βάση κιόλα αυτών των ε, θεμάτων και σε μια απλή βάση με τα άλλα θεσμικά όργανα για τη συνεργασία αυτή. Μπορώ να σας ε, αναφέρω ότι θυμάμαι ότι είχαμε εξαιρετική συνεργασία με το Συμβούλιο τότε και στο τέλος και φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την δημιουργία της συγκρότηση της όλα στην αρχή όπως μπορείτε να φανταστείτε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπösch, ε, στην αξιολόγησή σας ασκείτε επικρίσεις για το μικρό εύρος ε, των ερευνών της ε, Όλαφ που είναι 35% λέτε και θέλετε από 30% να το ανεβάσετε σε 50% τις ερευνητικές δραστηριότητες. Πώς οι δικές σας γνώσεις σε σχέση με τις έρευνες θα μπορέσουν ε, να αξιολογηθούν και να συνεισφέρουν. Διότι αυτό δεν απορρέει υποχρεωτικά από το δικό σας κουρίκουλουμ βείτε το δικό σας βιογραφικό. Δεν ήθελα να κάνω κάποια κριτική. θα πρέπει να βασιστώ στις εκθέσεις, γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν είμαι σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει όμως να πω ότι είναι ενδιαφέρον ότι από το 2004 μετά τη διεύρυνση μορονότι αυτό αύξησε το προσωπικό της Όλαβ η διάρκεια των ερευνών δεν μειώθηκε και δεν είχαμε και περισσότερες περιπτώσεις. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Είναι λογικό αυτό και αυτό θα πρέπει να αλλάξει όχι βεβαίως από σήμερα σε αύριο, γιατί ο διευθυντής της Όλαφ δεν μπορεί να πετάξει ανθρώπους έξω, αλλά πάνω σε μια πολύ ανθρώπινη βάση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. Περισσότεροι άνθρωποι δηλαδή να ασχοληθούν με την έρευνα περιπτώσεων. Αυτό αναμένεται από εμά. Ευχαριστώ. Κύριος Μπάτσιλης. Ευχαριστώ. Πραγματικά μου άρεσε η παρουσίασή σας. Σαφώς είπατε ότι για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις απαιτούνται αλλαγές. Και πραγματικά συμφωνώ μαζί σας σε ό,τι αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε διάφορους φορείς. Σε κάθε χώρα μέλος Υπάρχουν υπεύθυνοι φορείς που συμμετέχουν στην διερεύνηση περιπτώσεων απάτης. Για παράδειγμα, στη Λιθουανία έχουμε πέντε παρόμοιους ε, φορείς. Ε, το τμήμα ασφάλεια, τα τελωνία κτλ. Δεν έχουμε όμως ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αυτών των οργανώσεων και αυτό ικανοποιεί πάρα πολύ μερικούς παραβάτες. Στη χώρα μου συχνά συμβαίνει οι έρευνες να τραβάνε πάρα πολύ καιρό και το πρόβλημά μας είναι κατά πόσον είναι αντικειμενικές. Δεν νομίζετε ότι στις χώρες μέλη θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και θα πρέπει να δώσετε εντολή σε ένα και μοναδικό φορέα που θα είναι υπόλογος στην Όλαφ και θα είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση πληροφοριών για περιπτώσεις ε, απάτης. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στη μεταρρύθμιση της Όλαφ είναι μάλλον θέμα των εξωτερικών πτυχών της μεταρρύθμισης. Η νέα συνθήκη μας προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες, διότι στο παρελθόν, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, μόνον οι υπορισμένες προϋποθέσεις εάν δηλαδή η συνεργασία δεν καλύπτονται με την εθνική νομοθεσία, τότε ήταν δυνατό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Τώρα, με τη νέα συνθήκη, αυτό διαγράφηκε στη φράση και ο νέος διευθυντής είναι εκείνος που θα πρέπει να το διαπραγματευτεί με τα κράτη-μέλη. Διότι έχετε δει ότι υπάρχει κάποιο κενό. Και όταν μιλάμε για απάτη, για φοροδιαφυγή κτλ. Ε, το κενό αυτό, το έλλειμμα είναι επιζήμιο κυρίω όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Κύριο Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Μπόσ, γνωρίζετε φυσικά πολύ καλά αυτό τον Νίκο και αυτή την Επιτροπή. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Διαβλέπετε κάποιο κίνδυνο ή κάποια προβλήματα ε, επειδή υπήρξατε πολιτικό τόσο καιρό και τώρα αλλάζετε. Και δεν διαβλέπετε προβλήματα όσον αφορά αυτές τις σχέσεις. Μπορείτε να υποσχεθείτε ή μπορείτε να μας πείτε ότι θα είσαστε σκληρός απέναντι σε όλους μέσα στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι προηγούμενες σχέσεις σας, οι προηγούμενες εμπειρίες σας δεν πρόκειται να σας καθοδηγήσουν καθόλου στη συμπεριφορά σας και ότι θα λαμβάνετε τις αποφάσεις σας με αυστηρότητα αν κάποια στιγμή γίνεται ο νέος διευθυντής της Όλαφ. Thank Ευχαριστώ κύριε Σμίτ. Ίσως είναι το πιο ανοιχτό και το πιο διαφανές βιβλίο, ο πιο ανοιχτός που, ε, υποψήφιος που θα δείτε σήμερα και αύριο. Διότι αυτά τα οποία παρουσιάζουν μπορούν να είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Εάν πιστεύετε ότι ήμουν υπερβολικά ευγενή απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή του. Τελικά όμω, τα τρία βασικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να αποφασίσουν για το όνομα του νέου Γενικού Διευθυντή και για την Επιτροπή και τους Επιτρόπους. Το πρόσωπό μου δεν είναι κάτι το μυστικό. Είμαι γνωστός. Είναι γνωστό πώς θα συμπεριφερθώ. Και τελικά μπορεί κανεί να πει ότι υπάρχει μια περίοδος ηρεμίας εντωμεταξύ, εφόσον δεν είμαι ε, εν, ενεργός πολιτικός. Αν αυτό πιστεύετε ότι είναι εμπόδιο, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπέρς, είπατε ότι υπήρχε μια μη ισόρροπη σχέση όσον αφορά τα στοιχεία και τις δραστηριότητες τις οποίες κάνατε για τις έρευνες. Το 1 τρίτο είπατε ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνετε εσείς ώστε τουλάχιστον το ίμιση του χρόνου σας να αφιερώνετε σε ερευνητικές και διακριβωτικές δραστηριότητες και όχι ένα τρίτο αλλά το ίμιση τη εργασία τη Όλαφ να είναι εξεταστή, εξέταση. Ευχαριστώ. Θα uh, μιλήσω αγγλικά λοιπόν. Είπατε στην παρουσίασή σα ότι το 1 τρίτο των ερευνών μόνο το 1 τρίτο είναι έρευνε. Το 1 τρίτο. Και θέλετε να φροντίσετε να γίνει 50 και 50%. Ποιε είναι οι δραστηριότητε που θα επιβραδύνετε, που θα αλλάξετε, ώστε να φροντίσετε, ώστε θα φτάσετε σε αυτό το ποσοστό. Σε μια ισορροπία 50%-50% όσον αφορά ε, το προσωπικό, τις έρευνες και τη διοίκηση. Είναι δύσκολο να σας απαντήσω σήμερα. Η ιδέα είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό βοηθητικών υπηρεσιών και όχι επαρκή αριθμό ερευνητικών υπηρεσιών. Ο λόγος ύπαρξης της ΟΛΑΦ είναι η έρευνα που κάνει, διερεύνηση των προβλημάτων αυτών. Μπορείτε να κάνετε σεμινάρια για την πρόληψη απάτης κάθε εβδομάδα σε όλα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ικανοποιούνται ή όχι οι ενδιαφερόμενοι. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ε, ορισμένων ατόμων του προσωπικού. Το σημαντικό είναι να έχετε ένα σαφή στόχο και κατόπιν να δείτε πώς θα τον πραγματοποιήσετε το στόχο σας με τους σπόρους που διαθέτετε. Ευχαριστώ. Κύριε Μποκικόφσκι. Έχουμε σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με πολύ σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Μπέρς από πλευράς μου. Δεν έχω οποιαδήποτε επιφύλαξη ότι δεν θα είσαστε αντικειμενικός αν θα και όταν θα αναλαμβάνατε αυτό το αξίωμα. Είναι ένα θέμα πιστεύω προσωπικής ακεραιότητας και εντιμότητας ούτως ή άλλως και δεν θα ήταν κανένα πρόβλημα για σας τον ίδιο με το πολιτικό σας παρελθόν να υπομειστείτε τις ευθύνες του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ. Η ερώτησή μου αφορά το εξή θέμα. Κατανοώντας αυτό τώρα ότι οι δραστηριότητες της Όλαφ θα ενισχυθούν όσον αφορά τις έρευνες ε, κυρίως η καταπολέμηση της διαφθοράς ιδιαίτερα και η καταπολέμηση των απατών είναι πάρα πολύ σημαντικές υποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρουμε να έχουμε θεσμικά όργανα τα οποία θα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα και διοργανωμένα ώστε να μην είναι δυνατόν να υπάρχουν περιπτώσεις διαφθοράς και περιπτώσεις απατών και έτσι να δράσουμε και να δούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή συμφερόντων και από πλευρά των διαφορετικών θεσμικών οργάνων για την επίλυση προβλημάτων και για τον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πιο μεγάλη διαφάνεια, ένα μεγαλύτερο πιο ελεύθερο πλαίσιο και διαφάνεια που είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί. Ερωτώ λοιπόν, διερωτώ με, η Όλαφ δεν θα έπρεπε να στείλει, να αποστείλει ένα μήνυμα, να σηματοδοτήσει κάτι, ότι αυτή την κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Όλαφ ακριβώς, αυτή της διαφάνειας, να σηματοδοτηθεί αυτό και να δημιουργηθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα προωθήσουν ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά και όπου υπάρχει πρόβλημα να το αντιμετωπίζουμε θα έλεγα λοιπόν τέτοιοι μηχανισμοί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξεταστούν. Μπορείτε να μας πείτε τι έχετε υπόψη σας να κάνετε. Και εσείς και το Συμβούλιο και η Επιτροπή είστε εκείνοι που θα ορίσουν τους κανόνες. Ακόμα και ο ΛΑΕΦ πρέπει βεβαίως να λειτουργεί σεβόμενοι τους κανόνες, αλλά τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Και για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υπάρχει καλύτερη ενημερωτική πολιτική. Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο λιγμών και μόνοι σας μπορείτε να δείτε πόσες φορές έχετε ενημερωθεί από την Επιτροπή. Έχω την εντύπωση και άλλα θεσμικά όργανα δεν είναι πολύ ικανοποιημένα με το βαθμό ενημέρωσης. Συνεπώς αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί από πλευρά της ΟΛΑΦ. Και βεβαίω, όπω είδαμε στην περίπτωση τη Eurostat, υπάρχουν προβλήματα. Εάν κάποιο δεν έχει ενημερωθεί από την ΟΛΑΦ, όπω έγινε ε, στην περίπτωση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής, σε αυτή την πολύ σημαντική περίπτωση που θα θυμάστε. Λοιπόν, αυτή είναι μία απάντηση. Δεν είναι πλήρης απάντηση, αλλά είναι ένα σκέλος της απάντησης. Και δεσμεύομαι να ακολουθούσε μια πολύ ισχυρή ενημερωτική πολιτική, διότι αυτό είναι καθήκον του Γενικού Διευθυντή και κανενός άλλου. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην επαγγελματική σας εμπειρία, την πείρα σας. Σπουδάσατε κοινωνιολογία. Μετά είσαστε ε, σε κοινότητα που δραστηριοποιηθήκατε και μετά δράσατε ε, κομματικά για ένα χρόνο. Νομίζω είσαστε υπάλληλος ε, του Δήμου της κοινότητάς σας στα χαρακτηριστικά σας αναφέρετε, όπως είπε η κυρία Γκρέσλερ, ότι θα έπρεπε να καταδεικνύεται πείρα σε υψηλό αξίωμα σε σχέση με τη δικαιοσύνη, καθώς επίσης και επικεφαλής, ε, με την ιδιότητα επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας. Πού θα λέγατε ότι είναι ειδική η πείρα σας και εξαιρετική εμπειρία σας σε αυτά τα πεδία. Ευχαριστώ. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι ήμουν ο εισηγητής στη δημιουργία αυτού του θεσμού για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Βεβαίω εναπόκειται σε εσά να πείτε αν οι προσπάθειές μου στέφτηκαν από επιτυχία ή όχι. Εσείς είστε εκείνοι που μπορείτε να ψηφίσετε υπέρ ή κατά. Από την άλλη θα ήμουν ιδιαίτερα τυχής ε, αν δεν αντιμετωπίζετε ως πολιτικό. Βρίσκομαι ενώπιον σας ε, ως υποψήφιος για μια σημαντική θέση. Και θα πρέπει να πω ότι έχω κάνει αρκετές ε, δουλειές. Δεν, δεν εργάστηκα μόνο στην πόλη καταγωγής μου Εκεί ε, με προσέλαβαν γιατί είχα συγκεκριμένα προσόντα. Δεν νομίζω ότι η εικόνα που προβάλλεται εδώ σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς είναι σωστή. Νομίζω ότι τους πολιτικούς θα πρέπει να τους δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο κύριος Ολμέιερ. Η κυρία Ολμέιερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Μπέσου θα ήθελα μια ερώτηση να θέσω. Λιγότερο σε σχέση με το αν είναι κάποιος πολιτικός ή όχι και αν αυτό είναι προτέρημα ή μειονέκτημα, αλλά τα προσόντα θεωρώ ότι είναι σημαντικά ή τα προσόντα. Και σε αυτό θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Πρώτον, τι γίνεται, μια και επανειλημμένα και σε σημαντικό βαθμό έχουμε περιπτώσεις διαφθοράς. Πώς συγκεκριμένα, χειροπιαστά προτίθεστε εσείς να προωθήσετε την καταπολέμηση και την ποινική δίωξη των περιπτώσεων διαφθοράς, αλλά και για τις ερευνητικές δραστηριότητες. Ποιο κέντρο βάρους θα θέσετε που το έργο, την εργασία, το έργο της Όλαφ θα το προαγάγουν, θα το προωθήσουν. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω πώς η ανεξαρτησία της Όλαφ είναι ε, θέμα για σας. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό μέχρι στιγμή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόσβαση σε σχέση με στοιχεία είναι σαφέστερη παρότι εκτός. Πώς θα το λύσετε αυτό το θέμα αν βρισκόσαστε εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνει η Όλαφ στη θέση που είναι τώρα, δηλαδή στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρώτον, Πρώτο. Ενδεχομένως μπήκατε μέσα μετά από τη σύντομη παρουσίασή μου. Είπα ότι θέλω να αυξήσω τον αριθμό των ανακριτών από το 1 τρίτο στο 50% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων στην Όλαφ. Αυτό είναι ένα μέτρο, ένας για να είναι πιο σύντομε οι ανακρίσει και περισσότερο ικανοποιητικέ σε τελευταία ανάλυση. Δεύτερον, η Επιτροπή και ο εισηγητής ξέρει ότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσει τη μεταρρύθμιση της Όλαβε. Και αυτό είναι έργο των θεσμικών οργάνων. Ο διευθυντής της Όλαπ μπορεί να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Μπορεί να τίνει χείρα βοήθειας, θα λέγαμε. Αυτό είναι κάτι που έχει ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Μπαρόζο τόνισε ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για το μέλλον, δηλαδή η μεταρρύθμιση της Όλαφ. Εν ώψη της ε, ε, ε της θα μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει κάποια διαθεσμική όλα Όλα τα θεσμικά όργανα καλύπτονται από τη συνθήκη και είναι υπεύθυνα για την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θέμα, να ενδυναμώσουμε δηλαδή την ανεξαρτησία της όλα. Η ανεξαρτησία όμως δεν είναι κάτι που απειλήθηκε. Το Κοινοβούλιο αφιέρωσε μια ολόκληρη ημερίδα σε συνεργασία με διάφορα θεσμικά όργανα και όλοι τόνισαν ότι η ανεξαρτησία λειτουργήσε καλά θα λέγαμε υπό τους, ε, τον παρόντα κανονισμό. Η ιδέα μου, ναι, αυτή η διαθεσμική ρύθμιση που δεν ήταν δυνατή στο παρελθόν τώρα είναι δυνατή με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Βάουγκεν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε στην δήλωσή σας τονίσατε ιδιαίτερα το θέμα της ανάγκης μεταρρύθμισης της Όλαβα. Αν η Όλαφ είναι προς μεταρρύθμιση θα χρειαστεί ένα μια πάρα πολύ σωστή διαχείριση για να αλλάξουν οι μέθοδοι εργασίας και οι προτεραιότητες της οργάνωσης. Αναρωτιέμαι πώς θα το πετύχετε αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε ποιο θα είναι το στυλ διαχείρισης που θα υιοθετήσετε. Δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή αυτό. Υπάρχει μια δομή Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σε υψηλό επίπεδο και θα πρέπει κανεί να συνεργαστεί με το υπάρχον, εργατικό, ε, με το υπάρχον δυναμικό. Είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και φυσικές αλλαγέ. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν ή ε, άτομα που μετατάσσονται σε μία άλλη θέση εργασίας. Θα ήθελα στο μέτρο του δυνατού να καταστήσω άτομα από διάφορε υπηρεσίες με άτομα που ασχολούνται με τον τομέα της έρευνας. Εγώ δεν μιλάω για το 70% ή το 80%, λέω 50%. Το 50% θα πρέπει να ασχολούνται με τι έρευνε, με τι ανακρίσεις. Μία ιδέα που έχω στο μυαλό μου είναι ότι ο Γενικός Διευθυντής θα ήθελα να υπάρχει αυτός ο εθνικός δικαστής, η εθνική εισαγγελείς που θα έχουν άμεση σχέση με την Όλαφ και θα εργάζονται στο πλάι μου. Θα πρέπει να είναι άμεση σύμβουλη του Γενικού Διευθυντή. Είναι σαφές λοιπόν ότι κάθε περίπτωση που φτάνει στο δικαστήριο της μίας ή της άλλης χώρας θα πρέπει να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες. Αυτές είναι δύο ιδέες Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πέρσου. Την εξή ερώτηση πρέπει να ομολογήσετε στην υποψηφιότητα σας είπατε ότι οι ερευνητικέ δραστηριότητες της Όλαφ είναι το πιο σημαντικό για σας τον ίδιο. Και εγώ προσωπικά είχα την πείρα, την εμπειρία ότι με μια προσωπική τέτοια, ας το πω έτσι, αναφορά για την Όλαφ που αφορά ανταγωνιστή σας υπό αυτό το πρίσμα βρίσκω ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό ως μέσον. Πώς μπορείτε εσείς για μένα προσωπικά να με διασφαλίσετε, να μου διασφαλίσετε ότι θα είσαστε πραγματικά ανεξάρτητος ως Γενικός Διευθυντής της Όλαφ στο μέλλον. Ευχαριστώ. Again, Herr Ehrenhauser, I ask you to ε, ζήτησα να με δείτε ως υποψήφιο για αυτή τη θέση. Εσείς μιλάτε για πολιτικές πτυχές. Εγώ σας λέω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν ξέρω αν ποτέ ε, απευθυνθήκατε στην Όλαφ. Η Όλαφ δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε για να, για να είναι ένας φορέας όπου αποτείνεται κανείς εάν υπάρχει κάποια ύποπτη κατάσταση. Και τότε ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να αποφασίσει αν θα γίνουν έρευνες ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής κάνει έρευνες. Αυτό είναι το θέμα μας. Επειδή έχουμε άλλα 10 λεπτά στη διάθεσή μας, ας ακούσουμε μερικές ερωτήσεις ακόμα. Κυρία Γκρέσ, παρακαλώ. Εγώ πάλι, εντάξει. Να ξεκινήσω πάλι από την αρχή λοιπόν. Εντάξει, πολύ ωραία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτόν τον αυξημένο αριθμό των ε, ε, στελεχών στις έρευνες από 35% σε 50% δεν είναι ότι είναι αδρανείς και δεν κάνουν τίποτα. Είναι, ας το πω έτσι, ε, δραστηριοποιούνται για την ε, διερεύνηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από 35% να πάτε στα 50% για ερευνητικές δραστηριότητες είναι ένα σημαντικό μέτρο. Από πού θα αντλήσετε προσωπικό και ποιο έργο είναι εκείνο το οποίο θα εγκαταλείψουν αυτοί που θα ασχοληθούν με τις έρευνες. Quite. Είναι δύσκολο να σας απαντήσω με, με δύο λόγια. Από πλευράς μου υπάρχει δέσμευση. Αυτός είναι ένας στόχος. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αντικατασταθούν από κάποιον. Αυτή είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνω. Εάν πιστεύετε ότι ότι η Όλαφ διοικείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τότε ενδεχομένως υπάρχουν πολύ καλύτεροι υποψήφοι από μένα. Εγώ θα προσπαθήσω γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο για βελτίωση. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ετοιμότητα, μεγαλύτερη διάθεση των ε, εργαζομένων. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με έναν ξεκάθαρο στόχο και ο στόχος αφορά τις έρευνες και όλα τα άλλα έπονται. Ξέρω ποια είναι η δουλειά της Όλαβ. Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι τομείς ε, αρμοδιότητάς της, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές και αυτό ακριβώς έκανα την παρουσίασή μου ότι δεν θα ήθελα να καλλιεργήσω προσδοκίες αν δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι πόροι. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε πάνω σε κάτι. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι αποδεκτό αυτό. Καταλαβαίνω την Επιτροπή, καταλαβαίνω τους ενδιαφερόμενους ε, που μας λένε ότι έχετε ανοιχτές περιπτώσεις πολλά χρόνια. θα πρέπει κανείς να αναλάβει την ευθύνη. Να πει ότι θα βάλουμε τέλος ορισμένες περιπτώσεις, θα τις κλείσουμε, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις. Γκέιερ. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα για άλλη μια φορά είναι τα προσωπικά κίνητρα που έχετε. Έχουμε το θέμα των προσόντων το οποίο αναφέραμε πιο πριν από πλευρά σας. Ξέρω από προφορικές και προσωπικές συζητήσεις που είχαμε σε σχέση με την κατάσταση που είναι σαφής για σένα. Θα ήμουν ευγνώμων όμως αν εξηγούσε στα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής πού είναι το, η ικανοποίησή σου, ποια είναι η ικανοποίησή σου που σε οδήγησε στο να υποβάλεις υποψηφιότητα για αυτό το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή της Όλου. Uh, το είπα και στην αρχή. Ο λόγος είναι τραγικός. Οφείλεται στο θάνατο του κυρίου Γκρούνερ. Ε, δεν είχε συμβεί ε, αυτό το ατυχές συμβάν, δεν θα υπήρχαν υποψηφιότητε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που προσπάθησα να καταστήσω σαφές προτεραιότητά μου ήταν να προχωρήσουν τα πράγματα στον τομέα της καταπολέμησης των απατών στην Ένωση. Όλοι λένε χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση της όλα. Όχι ο μόνο ο πρόεδρος Μπαρόσο, αλλά και άλλοι. Πίστεψα λοιπόν ότι θα μπορούσα να συμβάλλω με έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Είμαι έμπειρος Βεβαίω, εσείς είστε εκείνοι που θα αποφασίσετε εάν στάθηκα πετυχημένος ή όχι. Αλλά είμαι σίγουρο ότι θα μπορούσα να συμβάλλω σε μία ε, μεταρρυθμισμένη όλα. Εσείς ως πολιτικοί θα μπορούσατε να μου δώσετε την απαραίτητη δύναμη. Αλλά θέλω μία χείρα βοηθείας και αυτό θα ήθελα για τα επόμενα ε, πέντε χρόνια. Η τελευταία ερώτηση, συνάδελφος Κόστιγκερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Από την υποψηφιότητά σας βλέπουμε ότι η Όλαφ ως διαθεσμικό όργανο θέλετε να λειτουργήσει και κυρίως για την ανεξαρτησία της ε, που πρέπει να διασφαλιστεί και με τη συμφωνία των θεσμικών οργάνων ε, για τις δραστηριότητες σας Ποια είναι τα προτερήματα και μειονεκτήματα θεωρείτε εσείς για την Όλαφ αν παραμένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι λέτε. Στην αρχή το 98, Το Κοινοβούλιο διατύπωσε μια, συνέταξε μια έκθεση που αφορούσε τη μεταρρύθμιση της Σούκλα. Η αρχική ιδέα του σώματος ήταν να υπάρχει μια διαθεσμική όλα. Αυτή ήταν η ιδέα τους και πιστεύω ότι θα ήταν ε, ενδιαφέρον να γίνει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε να παρετηθεί η Επιτροπή και οι δυνατότητες που είχαμε ήταν περιορισμένες. Η δυνατότητα που είχαμε ήταν να, να προσαρτήσουμε την Όλαφ με όλες τις, τις αρμοδιότητες είτε στο ελεγκτικό συνέδριο που δεν το ήθελε είτε στην Επιτροπή. Ήταν λοιπόν κάτι πολύ λογικό το ότι καταλήξαμε θα έλεγα σε αυτό το υβριδικό κατασκεύασμα. Αν μπορούμε όμως να το αλλάξουμε και αν υπάρχει πολιτική βούληση να το αλλάξουμε, θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να βοηθήσω σε αυτό. Αυτή δεν είναι καινούργια ιδέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Έρμπερτ Βός για την ακρόαση. Ευχαριστώ. Γεια σας. no está, no sono contento. Allora, diamo, okay. diamo uh, la parola adesso al secondo. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον δεύτερο υποψήφιο, στον κύριο Τιερή Κρετέμ. Ο κύριος Τιερή Κρετέ έχει πέντε λεπτά στη διάθεσή του για να μας παρουσιάσει την υποψηφιότητά του. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, καταρχήν θα ήθελα να σας πω πόσο μεγάλη τιμή αισθάνομαι που βρίσκομαι εδώ ενώπιον των εκπροσώπων των πολιτών. Πρώτα απ' όλα υπήρξα πρακτικός ε, εφαρμογή, ε, στο επάγγελμά μου και ένας ερευνητής. Επί 18 έτη υπήρξα ε, το θέμα ήταν, ήμουν μέλο των διοκτικών αρχών κατά του ξεπλήματο χρήματο και τη διεθνού απάτης. Παρουσιάζομαι με τις επιτυχίες που είχα στις μεγάλες δίκες, με μεγάλη απήχηση στον οικονομικό τομέα στη Γαλλία. Παρουσιάζομαι επίση με τα διάφορα λειτουργήματα που είχα αναλάβει στην Όλαφ από το 2001. Έρευνε στον τομέα των ε, τελωνίων, ε, απευθεία δαπάνε, εξωτερικέ ενισχύσει, εσωτερικέ έρευνε και όπου ή απάντοτε επιτυχία. Παρουσιάζουμε λοιπόν και μόλι την πανεπιστημιακή μου εργασία για το οργανωμένο έγκλημα και ε, την παγκόσμια εγκληματολογία. Θα ήθελα η Όλαφ να γίνει ένα κέντρο αριστεία. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι πρέπει να τοποθετήσουμε πάλι την Όλαφ στην κεντρική τη δραστηριότητα, οι έρευνε και τι λειτουργικέ δραστηριότητε ε, για να εξυπηρετούν την αναδιοργάνωση τη Όλαφ. Δεύτερον, πρέπει να εστιάζει τη προσοχή τη στι πιο περίπλοκε και δύσκολε περιπτώσει, εκεί όπου προσφέρει μια προστιθέμενη αξία και ένα νόημα. Τρίτον, η Όλαφ ε, ε, παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των πολιτικών πρόληψης της Επιτροπής με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών. Τέταρτον, είμαι αποφασισμένος να αντιμετωπίσω το πρόβλημα της διάρκειας των ερευνών από τρεις απόψεις. να θέσουμε σε νέα βάση τις λειτουργικές δραστηριότητες, το είπα ήδη, με την βελτίωση των μεθόδων εργασία και την καλύτερη επιλογή των περιπτώσεων. Πέμπτον, θα αναπτύξω τη συνεργασία με τους θεσμούς, τα κράτη-μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς Έξι, και αυτό είναι σημαντικό, η ΟΛΑΦ πρέπει να είναι ε, η υπηρεσία της νομιμότητας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα το συνοψίσω ως εξή. Αποτελέσματα και δίκαιη δίκη. Τέταρτο, έρχομαι τώρα στην εξαρτησία. Το χειρότερο για μια υπηρεσία ερευνών είναι να μην προσανατολίζονται οι, προ... οι δραστηριότητέ του, να χειραγωγούνται για να θίξουν ένα άτομο, ένα θεσμό. Η ανεξαρτησία είναι η εγγύηση τη ουδετερότητα και της αντικειμενικότητας των συμπερασμάτων. Χάρη στην εμπειρία μου των 30 ετών μιας ε, διαφοροποιημένης επαγγελματικής ζωής, ε, βασίζω την ανεξαρτησία στην ε, ικανότητα να αντιμετωπίσει κανείς τα διακυβεύματα. Τέλος, για μένα η ανεξαρτησία δεν πρέπει να γίνεται μεμονωμένα. Γιατί ένα άτομο σε απομόνωση δεν προσφέρει τίποτα το χρήσιμο. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι δεν είμαι ένα άτομο που εφαρμόζει τα πράγματα. Είμαι και οργανωτής. Έχω ε, την αίσθηση της καινοτομία ε, και της ηγεσία. Είμαι διπλο, έχω διπλωμάτης, ανοιχτός, ευέλικτος. Έχω σχέση εμπιστοσύνη με τους συναδέλφους μου. Γνωρίζω το περιβάλλον όπου εξελίσσεται η ΟΛΑΦ νομίζω ότι είμαι σε θέση να εξασφαλίσω και τη συνέχεια της υπηρεσίας και να της επιφέρω τις αναγκαίες αλλαγές για να αντιμετωπίσει το μέλλον. Με δύο λόγια, δεν ζητώ μόνο μια επαγγελματική εμπειρία. Νομίζω ότι μπορώ να αναλάβω την ευθύνη του διευθυντή τη ΟΛΑΦ, επειδή έχω την ικανότητα να παίρνω αποφάσει σε περίπλοκε και αβέβαιε καταστάσει. Καταλήγω αυτή τη σύντομη παρουσίαση μιλώντα για το μέλλον πρέπει να δίνουμε λύσεις στα άμεσα προβλήματα της Όλαφ για να προετοιμαστεί στις μελλοντικές αλλαγές στο χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Να λειτουργήσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ε, τις αλλαγές που θα απαιτήσει αυτό το τομέα με την Eurojust, με την Europol και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η υπηρεσία έχει συγκεκριμένες εμπειρίες διεθνούς συνεργασίες εδώ και χρόνια. Είναι σε θέση να προτείνει μια τεχνογνωσία μοναδική ώστε να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση. Ε, βραχυχρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάσουμε αυτό το όραμα μέσω και μακροπρόθεσμα που παραπέμπει σε μεγάλες μελλοντικές αλλαγέ και θα τοποθετήσει την Ελλάδα σε ένα κέντρο ω ένα απαραίτητο εταίρο μεταξύ των μεγάλων διεθνών ερευνητικών υπηρεσιών. Θέλω να σας πω όλα αυτά προκαταρτικά. Θα ολοκληρώσω όταν θα διευκρινίσω ότι στους θεσμούς ε, θα προσφέρω τη μεγάλη μου συνεισφορά. Η Επιτροπή σα και το Κοινοβούλιο. Πέραν από το σεβασμό που έχω για σας, πάντοτε μπορούν να στηρίζονται στην ευρύτερη συνεργασία μου και στην ανταλλαγή εξπεριών και επειδή γνωρίζω τη σημασία που έχει η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτή την υπηρεσία. Ευχαριστώ. Grazie. Onorevole Ja, vielen Dank für die σε ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Γκρέστερ, για την εντυπωσιακή παρουσίαση. Είσαστε ο υποψήφιο με την πιο συγκεκριμένη και ευρεία πείρα και εμπειρία όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και το δικαστικό επίπεδο επαγγελματικά. Μετά από δέκα μήνες ε, που ε, περάσατε, είσαστε εκείνος ο οποίος είσαστε ο πιο κατάλληλος άμεσα να ηγηθείτε της ε, Όλαφ. Και γνωρίζετε το αξίωμα με τα προτερήματα και τα ισχυρά του σημεία και τα αδύναμα σημεία του. Είσαστε επί αρκετό διάστημα σε αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό το μήνυμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας πείσει. Είσαστε μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Ποια είναι τα τρία άμεσα μέτρα τα οποία εσείς ως πιο κατεπήγοντα θα προτείνετε να υιοθετηθούν. Πρώτα μέτρα τα οποία θα ήθελα να προτείνω ε, στην ΟΛΑΦ έχουν σχέση με τη διάρκεια των υποθέσεων, το οποίο σημαίνει ότι πιθανόν θα πρέπει να υπάρξει αναδιοργάνωση. Επειδή πρέπει ε, να χρησιμοποιούνται οι πόροι εκεί που χρειάζονται. Υπάρχουν ίσως επικαλύψεις στην ΟΛΑΦ και απαιτείται καλύτερη κατανομή των μέσων που διαθέτουμε. Αυτό θα είναι το πρώτο μου μέτρο. Δεύτερον, θα, όπως και τώρα ως διευθυντής, θα δώσω προσοχή στην αποτελεσματικότητα των ερευνών μας. Το ανέφερα στην ομιλία μου. Είπα ότι η επιθυμία μου είναι, πώς να το πω, να εστιαζόμαστε στις πραγματικές υποθέσεις. Εκεί υπάρχει πραγματική απάτη. Καλύτερη επιλογή των υποθέσεων. Αυτό είναι καταλητικό για την αποτελεσματικότητα. Το τελευταίο έχει σχέση με το ρεαλισμό. Πρέπει να έχουμε μια σωστή μεθοδολογία Πρέπει να βελτιώσουμε τη μεθοδολογία μας. Πολλά πρέπει να γίνουν εκεί. Και σκοπεύω το ταχύτερο δυνατόν να συγκροτήσω την απαραίτητη ομάδα εργασίας. Γκέια. Γκέια, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Στην Όλαφ δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα ότι πώς να το πω, οι έρευνες ε, δεν είναι πλήρως τελεχωμένες και ότι έτσι οι περιπτώσεις είναι πιο χρονοβόρες ε, και δεν μπορούν να καλυφθούν και να επεξεργαστούν όπως ε, θέλουμε. Η δεύτερη ανησυχία που έχουμε είναι η εθνική συνέχεια που δίνεται, national follow-up. Ερώτησή μου, ποιες είναι οι δικές σας απόψεις ώστε συγκεκριμένα να αναλαμβάνετε ποινική δίωξη από τα κράτη και να βελτιωθεί αυτή η πτυχή. Ευχαριστώ. Όταν κάνω αναφορά στις συνθήκες, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να μοιραστούμε τι ευθύνε με τις χώρες μέλη. βασικό ρόλο ε, τη Όλαβ είναι να δημιουργήσει τι προϋποθέσεις καλύτερη ε, συνεργασία με τι χώρες μέλη. Σε ό,τι αφορά το δικαστικό κλάδο είναι το ίδιο πράγμα. Στην Όλαβ θα πρέπει να βελτιώσουμε Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει πολύ περιθώριο για βελτίωση θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τις πληροφορίες στο δικαστικό κλάδο. Γιατί όταν μεταφέρει κανείς ένα ημικατεργασμένο προϊόν, τότε ο δικαστικός κλάδος θα πρέπει να επιληθεί. Στην όλα, λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να δώσουμε στο δικαστικό κλάδο των χωρών μελών καλύτερο προϊόν. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πιστεύω. Για παράδειγμα, θα ήθελα να δημιουργηθεί μια καλύτερη ομάδα μονάδων για την παροχή νομικών ε, συμβουλών από την άποψη την κοινοτική αλλά και για την υποβολή διαμαρτυριών. Δηλαδή να είμαστε ένας πυλώνας πραγματογνωμοσύνης που χρειάζεται για να να μεταφέρουμε ορισμένα στοιχεία στι εθνικέ αρχέ και κυρίω στι δικαστικέ αρχέ μια χώρα μέλου. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να τονίσω Βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα με το δικαστικό κλάδο. Γι' αυτό το λόγο επιμένω σε ό,τι αφορά την δυνατότητά μας να δημιουργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και για να γίνουμε αποδεκτοί από τους συναδέλφους μας στις χώρες μέλη. επειδή λείπει ο κύριος Λιβέλη, κυρία Γκρέσ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η μεταρρύθμιση της ΣΟΛΑΦ επίκειται και πάλι τίθεται το θέμα της ανεξαρτησίας του Γενικού Διευθυντή που είναι πολύ σημαντική κατά τη δική μας άποψη. Εδώ και δέκα χρόνια η Επιτροπή Επιτήρησης δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Νομίζω ε, όμως ότι πρέπει, πώς βλέπετε την αντισκρατησία της ΟΛΑΦ και πώς πιστεύετε ότι θα ενεργήσετε στα πλαίσια της Επιτροπής Παρακολούθησης εάν διακυβεύεται ανεξαρτησία, διότι ως ε, αξιωματούχος Επιτροπής ο Γενικός Διευθυντής έχει δυσκολίες να στραφεί κατά του ίδιου του θεσμού του. Τι συμβαίνει λοιπόν με την ανεξαρτησία και τις σχετικές διαδικασίες για να διαφυλάξετε την ανεξαρτησία. Ένα ουσιαστικό θέμα είναι αυτό και πολύ ευαίσθητο. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με κάτι άλλο. Ευθύ εξ αρχή θα ήθελα να σας μιλήσω ότι για να είναι κανείς ανεξάρτητος σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε θέση να είναι ουδέτερος και αντικειμενικός στα συμπεράσματα μιας έρευνας. Επίσης σημαίνει να προχωρήσει κανείς αρκετά όσους επιτρέπουν όμως τα τεκμήρια. Λοιπόν, μιλώ για γεγονότα και για τίποτε άλλο. Πιστεύω όμως ότι για να υπάρχει ανεξαρτησία χρειάζονται να πληρούνται ορισμένε προποθέσει. Πιστεύω ότι πρέπει να βασίζεται κανεί και στην εμπειρία. Το ανέφερα στην εισαγωγή μου ότι η εμπειρία είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό υπό την έννοια ότι θα πρέπει να δείτε Πού ε, διακυβεύεται η ανεξαρτησία σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να το μάθετε από την εμπειρία σας. Και επίσης πρέπει να είστε πολύ προσεκτικός. Αυτή είναι η προσέγγιση μου λοιπόν. Δεν εξαρτάται μόνο από τα άτομα, αλλά εξαρτάται και από το νομικό περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα πρέπει να αναφέρετε. Και πάλι η ανεξαρτησία δεν είναι ένα προνόμιο. Για μένα η ανεξαρτησία είναι ένα καθήκον το οποίο θα υπομίζεται ο διευθυντής τη ΟΛΑΦ. Σημαίνει ότι δεν είσαι ελεύθερος να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, αλλά θα πρέπει να, ε, ε, ε, να είσαι υπόλογο, υπόλογο σε εσά στην Επιτροπή. Και για να έλθω τώρα στο θέμα που θίξατε, το οποίο αφορά το πρόβλημα των προβλημάτων με την ιεραρχία στην Επιτροπή, επειδή αυτό αναφέρατε και πάλι θα πρέπει να βρίσκουμε στη σωστή θέση ενώπιον των ευθυνών μου. Τη στιγμή που έχετε ε, αναλάβει μια αποστολή πρέπει να την εκπληρώσετε. Και έτσι το, τα βλέπω. Εάν χρειάζεται τα πράγματα να τα, δει, να τα, να τα τεθούν υπόψη της Εποπτικής Επιτροπής ή αλλού, θα το κάνω, θα το κάνω. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, κύριε pretendentė. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφι. συμφωνούμε όλοι ότι έχετε μεγάλη πείρα στον τομέα των ερευνών. Και αυτό είναι αυτό που χρειάζεται αυτός ο φορέας. Αναφερθήκατε στην βούληση που έχετε. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν θα είναι πάντοτε δυνατόν να εφαρμόσετε αυτά που έχετε στο νου σας, γιατί το δυναμικό που έχετε, το ανθρώπινο δυναμικό είναι περιορισμένο. Και υπάρχουν και οικονομικοί περιορισμοί. Παρ' όλα αυτά χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις καλές σας προθέσεις. Είπατε ότι θα προσεπαθήσετε να κάνετε μια καλύτερη επιλογή των περιπτώσεων. Νομίζω ότι είναι καθαρά υποκειμενικό όμω αυτό το θέμα. Κάτι άλλο που είπατε αναφερόταν στα διαρθρωτικά ταμεία. Έχουμε πολλά προβλήματα με τα διαρθρωτικά ταμεία. Πάνω από το 50% όσων ασχολούνται με το τομέα των ερευνών λένε ότι το πρόβλημα με τα διαρθρωτικά ταμεία είναι η πολύπλοκη διαδικασία επιλογής. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας, θα επιθυμούσαμε να σας βοηθήσουμε με όλες τις ε, δραστηριότητες που αφορούν, τις ενέργειες που αφορούν τα διαθωτικά ταμεία. Έχετε ιδέα όμως τι σκοπεύετε να κάνετε με τα διαθωτικά ταμεία. Έχετε κάποιο όραμα μπροστά σας. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των περιπτώσεων, γιατί από την ερώτησή σας, από μόνο αυτό το μέρος, πιστεύω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό θέμα για την Όλαφ. Η Όλαφ θα πρέπει να είναι ένας ανακριτικός, ένας ερευνητικός, ε, ανακριτικός φορέας, ο οποίος θα πρέπει να ξεχωρίζει ορισμένες περιπτώσεις. Αν πάρω το θέμα των διορθωτικών ταμείων, είναι κοινά με τις χώρες μέλη. Υπάρχει λοιπόν διπλή ε, ευθύνη και της ε, ε, Επιτροπής και των χωρών μελών να κάνουν ό,τι καλύτερο. Είναι αρκετά σαφές για μένα ότι όταν έχουμε να κάνουμε με οργανωμένο έκλημα πολύ συχνά μιλάμε για ατασταλίες, ενώ θα πρέπει να μιλάμε για διαφθορά ή για πάτες. Αυτά είναι προσχεδιασμένα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια καλύτερη επιλογή των περιπτώσεων. Πιστεύω επίσης ότι με βάση τα αποτελέσματα των επιλεγμένων ε, περιπτώσεων θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτρεπτικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Το άλλο που είπατε είναι πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πιστεύω ότι από τις έρευνες που ήδη έχουν διεξαχθεί θα μπορούσαμε να πάρουμε πολλά διδάγματα. Και αν ξέρουμε να τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα διδάγματα, δίχως άλλο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Η Επιτροπή είπε και συμφωνώ γιατί είναι και δική μου πεποίθηση ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την κατάληξη, από τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. Πρόσφατα στην Όλαφ είχαμε μία περίπτωση όπου μπορέσαμε να κάνουμε μία ενδελεχέστατη ανάλυση και με βάση αυτό η Επιτροπή και θα μπορούσε να ισχύσει και για τις χώρες μέλη θα μπορούσε να μάθει πάρα πολλά για να ε, δεν είναι τα πάντα στα χέρια της Όλαφα, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες στους εταίρους μας και στους ενδιαφερόμενους για να μπορέσουν να διορθώσουν το σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κρετέν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε την απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως υψηλό τέλεχος στον τομέα του management. Ε, ανήκατε κάποτε σε κάποια επαγγελματική οργάνωση. Σε ποια και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελευταία ερώτηση. είχατε εμπλακεί σε μία καταγγελία για μόμπινγκ. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πού αναφέρεται αυτή η καταγγελία. Ωραία, να μιλήσω αγγλικά. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε. Σε ό,τι αφορά το, την ένταξή μου σε ένα σωματείο ε, το παρελθόν ε, είχα ορισμένες επαφές με ένα σωματείο, με ένα σύλλογο δικαστών στη Γαλλία. Πέρα από αυτό τίποτα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, δεν καταλαβαίνω που αναφέρεστε. Μήπως θα μπορούσατε να γίνετε περισσότερο ακριβείς για πέστε μου. Θα μιλήσω και πιο αργά για να μπορέσουν να μεταφράσουν οι διερμηνείς. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχετε την απαιτούμενη εμπειρία των πέντε ετών σε υψηλόβαθμη θέση και αν ναι, πού και τι ρόλο είχατε. Δεύτερον, αν ανήκατε σε επαγγελματικά σωματεία και αν ναι για πόσο χρόνο. Μιλήσατε για ένα συνδικάτο. Θα ήθελα να γνωρίζω τι ήταν, ένα σωματείο, ένα συνδικάτο, τι. Τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν έχετε εμπλακεί σε μία καταγγελία για μόμπινγκ από πλευράς ενός ανώτατου ε, οικονομικού ε, ε, αξιωματούχου στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας το ε, να γίνετε πιο σαφείς. Ναι, ναι, υπήρξα. Αναφέρεστε σε ένα, με μια οργάνωση, σε ένα σωματείο. Ναι, ήμουν στην επαγγελματική οργάνωση των δικαστών. Ναι, αναφέρω ότι είχα εμπειρία στον τομέα του management ε, για διάστημα μεγαλύτερο το 5 ετών. Για παράδειγμα, ήμουν ε, εισαγγελέα ε, στη Γαλλία για 6,5 χρόνια. Ήμουν υπεύθυνο για τον προπολογισμό και για μια σειρά από πράγματα που δεν είναι η καθημερινή εργασία του. Ε, εισαγγελέα, αλλά είναι θέμα διαχείρισης. Όταν έφτασα στο δικαστήριο, το δικαστήριο αυτό έπιασε με ένα δικαστήριο του 19ου αιώνα. Όταν έφυγα το 1993 είχε γίνει ένα δικαστήριο του 21ου αιώνα, απόλυτα εξυγχρονισμένο. Έκανα πολλές έρευνες. Χρησιμοποίησα τον προπολογισμό για να βελτιώσω τις συνθήκες εργασίας. Αναφερθήκατε σε ένα, μια διαμαρτυρία. Ναι, ναι, πρόσφατα κάποιος διαμαρτυρήθηκε από έναν υπεύθυνο της οικονομικής αστυνομίας την Guardia di Finanza και ζήτησε την προστασία του άρθρου 22. Από ό,τι γνωρίζω είναι κάτι που είναι ακόμα υπό εξέταση ασχολούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Στάις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κρετέν γνωρίζει ότι εμείς ως βουλευτές πολύ συχνά συναντώμεθα με υπεύθυνους της Όλαβ. Θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια είχα την εντύπωση είχα την εντύπωση και είχα για πληροφορίες ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στη λειτουργία της Όλαφ και ότι μερικές φορές μιλάμε για τη δημιουργία ε, ομάδων και ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στα πλαίσια της Όλαφ. Αυτό είναι κάτι που επιβραδύνει τις εργασίες της Όλαφ και επιβραδύνει και την, ε, τον όλο μηχαν, τη λειτουργία όλου του μηχανισμού. Θα ήθελα να μου πείτε, επιβεβαιώνετε αυτή την ανάλυση. Επιβεβαιώνετε ότι όντως έχει έτσι αυτή η κατάσταση. Και αν ναι, πώς κατά την άποψή σας αυτές οι συγκρούσεις μέσα στο εσωτερικό της όλα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν ή να επιληθούν με τη δική σας συμβολή ως Γενικού Διευθυντή. Ε, είναι αλήθεια. Αναφερθήκατε στη λέξη ομάδες. Δεν θα τις αποκαλούσα ε, έτσι. Είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ε, απόψεις. Υπάρχει μια σύγκρουση. Ναι, θα μπορούσε να μεταβληθεί σε σύγκρουση. Σε τελευταία ανάλυση όμως δεν είναι είναι ένας ε, διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ορισμένων πραγμάτων. Αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το να γνωρίζουν οι άνθρωποι σαφώς ποια είναι η αποστολή τους. Και μερικές φορές, φορές αυτά δεν τα γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν την αποστολή τους, δεν, γνωρίζουν τις μεθόδους εργασίας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η έρευνα για να στοχοθετηθεί κάποιος, στοχοποιηθεί κάποιος. Πώς θα μπορούσα όμως να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα εάν, ποτέ, εάν γίνω Γενικός διευθυντή. Για μένα τα πράγματα είναι μάλλον απλά σε αυτό το τομέα. Το πρώτο πράγμα είναι να μάθει κανείς να ακούει. Ποιο είναι το σημείο εκκίνησης για τις συγκρούσεις το σημείο κίνηση έχει σχέση με το γεγονό ότι οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ του. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε το πρόβλημα, να μιλήσουμε. Και αφού μιλήσουμε θα μάθουμε από αυτό και θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε από κοινού τη λύση. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να ε, πορευτώ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να διευκρινίσω σε αυτή τη φάση. Εάν υπάρχει πλήρης διχογνωμία μεταξύ δύο ατόμων, ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι επίκυνται αλλαγές στην Όλαφα. Εάν ε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ευτυχείς με τις αλλαγές, τότε αυτό δημιουργεί κάποια αντίδραση και πολλοί το, λένε, το ονομάζουν σύγκρουση. Δεν είναι σύγκρουση. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα και λόγω αυτών των βελτιώσεων οι άνθρωποι νιώθουν ανασφαλείς είναι εναπόκειται στην ε, διοίκηση και στον υπεύθυνο να εξασφαλίσει ότι όλα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πολλά και θα πρέπει να γνωρίσουμε προς τα πού προσανατολίζεται η Όλαφ και να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των συγκρούσεων και από τη μία πλευρά και των διαφορετικών προσεγγίσεων από την άλλη. Ευχαριστώ. Η ομάδα ICR υπάρχει ε, κάποιος εκπρόσωπος. Αν όχι, συνεχίζουμε. Κύριε, ε, ε, κύριε Ανδρεάς. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κρετά, μπορείτε να μας πείτε αν πιστεύετε ότι οι, οι καταδότες κατά κάποιο τρόπο είναι σημαντική ομάδα στις ερευνές σας και αν αυτή τη στιγμή ε, διερευνάτε τις ανώνυμες καταγγελίες. Whistleblowers are a tool disposal. είναι ένας ε, μηχανισμός ε, στη διάθεσή μας. Από στατιστική άποψη, θα σας πω, δεν έχουμε πολλούς καταδότες υπό τη στενή έννοια της ε, λέξης. Αλλά κάθε μέρα η ΟΛΑΦ έχει να κάνει με πολλές ανώνυμες καταγγελίες και λαμβάνουμε πολλές ανώνυμες καταγγελίες. Πληροφοριοδότες δηλαδή είναι αυτοί. Ναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Είναι πάντοτε πρόβλημα να ανακαλύψει κανείς την απάτη, διότι χωρίς ε, την ανείχνευση απάτη δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικό όταν μου δίνονται ανώνυμε πληροφορίε, διότι εκείνο που διακυβεύεται πολύ συχνά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πώ μπορώ εγώ να ελέγξω κατά πόσον μια κατηγορία, ένα υπενιγμό είναι αρκετά σοβαρή, εάν δεν ξέρω από πού προέρχεται, ποιο είναι ο πληροφοριώτη μου δηλαδή. Πολλέ φορέ έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και όπω γνωρίζετε, και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό πάρα πολύ, Τη στιγμή που λαμβάνουμε μια πληροφορία στην ΟΛΑΦ την αξιολογούμε, την εκτιμούμε για να δούμε κατά πόσον είναι αρκετά σοβαρή. Αν αυτή η υπόνοια δηλαδή είναι αρκετά βάσιμη. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα φάκελο. Και αυτή η δουλειά γίνεται πραγματικά ενδελεχώς. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι λαμβάνουμε πολλές ανώνυμες πληροφορίες και καταγγελίες καθημερινά. Αλλά και ε, άλλες καταγγελίες επώνυμες. Βεβαίως λαμβάνουμε και ανώνυμες. Τόσο, όσον αφορά τους πληροφοριοδότες, τους καταδότες, δεν έχουμε πολλούς. Ευχαριστώ, κύριο Στάις ήδη υπέβαλε εν μέρη το ερώτημά μου. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς ε, βλέπετε τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μονάδων και υπάρχουν ορισμένε αδυναμίε που μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά ήδη με καλύψατε. Λοιπόν, θα μπορούσα να σα ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να μα πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα που ένα συμπυρογνώμων όπω εσεί, που ήδη έζησε αυτή την οργάνωση, Πώ μπορείτε να εφαρμόσετε καλύτερα τι διαδικασίε πώ να βελτιώσετε την κατάσταση καλύτερα από έναν άλλον εξωτερικό υποψήφιο.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 πάντοτε δύσκολο να μιλήσει κανεί για τον εαυτό του. Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλω μία προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό συντονισμό, είναι σημαντικό. Υπάρχει έλλειψη εσωτερικού συντονισμού στην Όλαφ. Και η δική μου αίσθηση είναι ότι θα πρέπει να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε εκεί. Πριν να δώσω μία απάντηση στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, θα περάσω στο επόμενο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι δύο παράλληλα θέματα. Η Όλαφ είναι ένα πολύ σύνθετος φορέας. Αν κάποιος έρχεται από έξω θα του χρειαστεί αρκετός χρόνος πριν να τα καταλάβει όλα και να τα αφομοιώσει. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων, δεν είναι θέμα ευφυΐας, είναι καθαρά θέμα χρόνου. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι εγώ μπορώ να ξεκινήσω με ένα προσωπικό που το γνωρίζω. Ξέρω ποιος κάνει τι, ξέρω ποιος είναι ικανός σε κάθε τομέα. Ξέρω την ιστορία που έχει πίσω της η Όλαφα. Ξέρω το περιβάλλον. Ξέρω πολλές Τυχέ τη ε, ε, εργασία εκεί, γιατί έχω εργαστεί σε έξι διαφορετικού τομεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσα να ξεκινήσω από την πρώτη κιόλα μέρα. Ενδεχομένω υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ. Θα μπορούσατε να αναρωτηθείτε κατά πόσον εάν οριστώ γενικό ε, διευθυντή, τα πράγματα θα αλλάξουν ε, από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν τα άλλαξα μέχρι τώρα γιατί δεν ήμουν γενικός διευθυντή. Και γιατί άρχισα να κάνω μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν είναι ορατά. Έκανα όμω πολλά κατά τη διάρκεια τη ε, ε, εργασία μου. Έβαλα μία τάξη, έδωσα σαφεί οδηγίε ε, για τα χρονοδιαγράμματα. Κατέβαλα προσπάθειες για να γίνει ένας προγραμματισμός της εργασίας των ερευνητών, των ανακριτών. Έκανα πολλά σε μια προσπάθεια να βελτιώσω τις ε, ε, σχέσεις με άλλους φορείς. Για να επανέλθω τώρα σε μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις, αυτός είναι ένας από τους τρόπους για να ελαφρύνει κάπως το άχθος των ε, ανακρίσεων. Αυτό είναι μέρος του εσωτερικού συντονισμού. Λιμπεράσκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν κύριε Κρέτα, σας παρακολούθησα προσεκτικά και έχω την εξή εντύπωση που αποκόμισα. Δυναμική παρουσίασή σας, σίγουρα. Όμως, όμως, είσαστε στην όραφα, έχετε ε, επί αρκετό χρονικό διάστημα, έχουν υποβληθεί προτάσεις, αν έχουν υποβληθεί και έχουν ε, απορριφθεί, τότε τι γίνεται με τους όρους εργασίας ε, υπό τους οποίους λειτουργήσατε. Οι σκέψεις σας είναι ενδιαφέρουσες ε, σκέψεις. Όμως, από την άλλη πλευρά, η τελευταία σας απάντηση κάπως μας εξέπληξε. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το θέμα το, του πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί η Όλαφ και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα το δυναμικό και τις δυνατότητες και τις πληροφορίες που έχει. Ευχαριστώ. Η Όλαφ θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάκτηση των χρημάτων υπό τον όρο ότι θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες και δεν εξαρτούν σωστά οι έρευνες. Αναφέρατε το γεγονός ότι μοιάζω δυναμικός. Μπορώ να σας πω ότι όντω είμαι δυναμικό και μερικέ φορέ αυτό προξενεί τη δυσαρέσκεια τη συζύγου μου. Μερικέ φορέ απορρίφθηκαν οι προτάσει μου. Ένα παράδειγμα. Επέμενα για πολύ στην Όλαφ για να υπάρχει ένας κανόνας διαδικασίας πολύ πιο ε, ή ένας εσωτερικός κανονισμός που να είναι πολύ πιο λεπτομερής, να υποβάλλονται σαφείς προτάσεις. Όταν ε, είμαστε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δέχουμε ότι θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις. Θα πρέπει να καταλήγουμε όμως σε συμπεράσματα. Θα πρέπει να αποφασίζουμε κάθε φορά τι να κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που σας δίνει μία ιδέα. Αν τα πράγματα είναι σαφή σταθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τότε μπορούμε να έχουμε σαφεί κανόνε, σαφή συμπεριφορά, σαφεί προσανατολισμού. Κατά την άποψή μου είναι περισσότερο θέμα διαχείριση, περισσότερο θέμα προσανατολισμού. Δηλαδή το να χαράξουμε την πορεία μας και να κινηθούμε προς μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το ανέφερα στην αρχική μου παρέμβαση και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σαφές. Κινούμεθα έτσι, μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί έχουμε στην Όλαφ όλη την πραγματογνωμοσύνη. Ενδεχομένως μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Δεν χρησιμοποιήσαμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ερενάουζερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρκετά χρόνια εντωμεταξύ εργάζεστε στην Όλαφ. Θα θυμόσαστε την περίπτωση του Hans Martin Tiller του 2004 που είχε ξεκινήσει μια ερευνητική δραστηριότητα από πλευράς ε, Όλαφ και μια απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που είχε πει ότι είναι παραβίαση της ελευθερίας ε, της πληροφόρησης. Πώς ε, τώρα κάποια χρόνια μετά θα το αντιμετωπίζατε αυτό και πώς θα κρίνατε τη δράση της Όλαφ τότε. Ευχαριστώ. Πριν από λίγο αναφέρθηκα στην ανάγκη να κατανοήσουμε την ε, ιστορία της Όλαφ. Εγώ αποτέλεσα μέρος της ιστορίας αυτής. Για να μην μακρηγορώ θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Όλαφ έκανε λάθη. Κάναμε τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν ήταν ο σωστός. Αλλά από την νομική ε, άποψη δεν κάναμε λάθη, δεν κάναμε κάτι που ήταν λανθασμένο. Το πρόβλημα είναι ότι στην περίπτωση Τίλακ πολλά προέρχονται από έξω, αλλά ήταν από μέσα. Και ανοίξαμε την περίπτωση, την διερευνήσαμε και καταλήξαμε σε ένα συμπέρασμα, γραπτόσο. Και, όπως είναι υποχρεωτικό, στείλαμε τις πληροφορίες αυτές στο δικαστικό κλάδο στις ε, Βρυξέλλες. Ξέρετε ότι θεωρήθηκε ότι η στάση του δικαστικού σώματος Βρυξέλλες δεν ήταν σωστή. Ενδεχομένως θα έπρεπε να το είχαμε κάνει με διαφορετικό τρόπο είναι εύκολο να ξαναγράψει κανείς την ιστορία. Αυτό όμως είναι μέρος, κομμάτι της ιστορίας της Όλαφ. Δίχως άλλο, μέσα στην Όλαφ υπήρχαν φράξιες, υπήρχαν ομάδες που συγκρούονται η μία με την άλλη. Αυτοί, αυτές οι πληροφορίες βγήκαν και προς τα έξω. Αυτό είναι κάτι όμως που αφορά το παρελθόν και φαντάζομαι ότι δεν θα ξανασημειωθεί κάτι τέτοιο θα έλεγα ότι θα με απασχολήσουν πολύ αυτά τα θέματα γιατί έχουν σχέση με την ικανότητα της Όλαφ να μην αφήνει πληροφορίες να διαραίουν και με λάθος ε, τρόπο. Αλλά βεβαίω στον τομέα αυτό έχουμε όλο και λιγότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρετέν για την ακρόαση και συνεχίζουμε. siamo? Ξεκινάμε με την τρίτη ακρόαση, να καλωσορίσουμε τον κύριο Τζον Ντένοφ, στον οποίο θα ήθελα να δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το ότι προσκλήθηκα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρίσκομαι εδώ και έχω ευκαιρία να σας εκφράσω τις απόψεις μου για το μέλλον της ε, Όλαφ και για να το κάνω αυτό ουσιαστικά ξεκίνησα σε σχέση με το benchmarking που είναι η προστασία ακριβώς ε, των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω και κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό και φυσικά οι συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου είναι κάτι σημαντικό σε σχέση με το ίδιες τις ερευνητικές δραστηριότητες και τον νέο ρόλο της Εποπτικής Επιτροπής. Και δεύτερον, συγγνώμη, σαν ένα δεύτερο στοιχείο και με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μια σύντομη επισκόπηση που μας δείχνει ότι 87,5% είναι αντικείμενο ε, απατών, πολλαπλών απατών. Και το τέταρτο είναι οι δραστηριότητες ε, της Όλαφα δεν λαμβάνει υπόψη ακριβώ του κινδύνου σε σχέση με τον ε, προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι 33% των δραστηριοτήτων αφορά η ε, δράση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και σε σχέση με την ετήσια αυτή η έκθεση, τα στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι δεν έχουν οδηγηθεί πάρα πολλέ περιπτώσει σε ανάκτηση και έχουμε εδώ το θέμα των στατιστικών στοιχείων και όσον αφορά τον όγκο την, της ε, ε, ερευνητικής δραστηριότητας για αυτές τις περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες οι διαδικασίες. Σε κάποιες διαφάνειες λοιπόν και σε κάποιες ε, τέτοιες παρουσιάσεις θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά βραχυπρόθεσμα θα ήθελα να αποκατασταθεί η, α, ηρεμία και αποτελεσματικότητα και εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της συνέχειας συνέχεια, μια και ήταν ε, επί αρκετό διάστημα η, το, η Όλαφ χωρίς Γενικό Διευθυντή. Ζητώ 100 ημέρες, όχι τίποτα περισσότερο. 100 ημέρες για την έγκριση του σχεδίου λειτουργίας τη Όλαφ από πλευρά μου και μετά μπορούμε να στραφούμε στο έργο θα ήθελα να πω ότι πρέπει να επανέλθει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της η Όλαφ, προστασία των οικονομικών δραστηριοτήτων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εδώ και σε σχέση με την ανάκτηση ποσών να υπάρξει αντίστοιχη δράση. Θα ήθελα να επανεστιαστεί η Όλαφ στις εξωτερικές ε, ε, διακριβώσεις και εξετάσεις και αυτό θα ήταν ένα καλό μέσο, ένα καλό εργαλείο. Τούτου λεχθέντος γνωρίζουμε ότι το μονοπόλιο για τις εσωτερικές ε, εξεταστικές δραστηριότητες ε, και μάλιστα με ε, ελάχιστο, με μηδενικό ποσοστό ανοχής και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 44% των ανακτηθέντων ε, καταφέραμε να τα ανακτήσουμε μέσω συνεργασίας ε, και των κρατών μελών και αυτό πρέπει να αυξηθεί στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και την Eurojust, ε, με την Eurojust και την Europol και να προσπαθήσουμε να έχουμε ανταλλαγή απόψε, ε, στοιχείων, ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνεργασία αυτών των φυσικών από τη φύση τους εταίρους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετηθεί η εσωτερική δομή της Όλαφ, να έχουμε την ε, ανάλυση των δραστηριοτήτων και δεν χρειάζονται περισσότερα κονδύλια. Είναι επαρκές το πλαίσιο του προϋπολογισμού της Όλαφ για να καλυφθούν οι δραστηριότητες Έχω κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ε, μπορέσει να λειτουργήσει η αξιολόγηση περιπτώσεων, να έχουμε ένα ενιαίο σημείο επαφής και ε, ε, δασ δεσμών με τα κράτη-μέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών και τις ανταλλαγές στοιχείων με την Europol, Eurojust. Σε αυτή θα πρέπει να δούμε τον ρόλο το, σε σχέση με τις εξεταστικές δραστηριότητες και να δούμε 35% συνολικά των δραστηριοτήτων των στελεχών 35% αφιερώνονται μόνο στις ε, ερευνητικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής ε, θα πρέπει να έχει ανοιχτό πνεύμα για να συζητήσει το πλαίσιο, το εύρος των δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στις ε, εξεταστικές αυτές δράσεις της Όλαφ που πρέπει να προστατευθούν και να προαχθούν. Λοιπόν, από πλευράς ε, ε, αστυνομία στο Βέλγιο που ήμουν ε, επικεφαλής αρμόδιος επί δεκαετίες τώρα, σχεδόν ολοκληρώνω, ευχαριστώ. Έχω λοιπόν σημαντικό πλαίσιο παρακαταθήκη πείρας και νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω, διότι έχω και μια διαφορετική ε, γνώση του τι συμβαίνει στην ε, Όλαφ ε, μέσω των, της εμπειρίας μου και θα πρέπει να αναφερθώ σε σχέση με τις δραστηριότητές μου οι περισσότερες περιπτώσεις έρευνας περιπτώσεων διαφθοράς στο Βέλγιο είναι εκείνες που έχουμε παρακολουθήσει από κοινού με την Όλαφ και βέλτιστες πρακτικές που δείχνουν ότι αν δράσει κανείς άμεσα και αν συνεργαστεί κανείς από κοινού με τα κράτη-μέλη μπορεί να επιτύχει θετικά αποτέλεσμα. Μεταξύ 2008-2011 έχουμε προαγάγει ε, σημαντικές ε, αποφάσεις ε, με την συνεργασία όσον αφορά τις βελγικές ερευνητικές αρχές, πράγμα το οποίο ήταν θετικό. Ευχαριστώ. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάπως με τώρα πρέπει να πω. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει ένα ολόκληρο ε, κύμα αντιδράσεων διότι ε, είπατε μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που ε, θα είναι ευχάριστα εσωτερικές εξωτερικές εξεταστικές δραστηριότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάτι εδώ διότι έχουμε και το θέμα της αξιοπιστίας. Το δεύτερο σημείο, τι θα γίνει με την ίδια την Όλαφ. Η το ανοιχτό αυτό πλαίσιο, το οποίο εσείς ως Γενικός Διευθυντής θα θέλατε να πετύχετε για μια υπηρεσία και αν γινόταν ακριβώς η, η Όλαφ μια τέτοια υπηρεσία, μια τέτοια οργάνωση, είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να παραμείνει η Όλαφ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να έχουμε έναν γενικό διευθυντή που θέλει το αντίθετο αυτού που επιθυμούμε εμείς, πώς μπορεί να το δεχτούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς μπορεί αυτό να συνάδει με τους δικούς μας στόχους, πώς θα σας ε, εκλέξουμε εμείς. Νομίζω το πρώτο είναι ότι υπήρξε κάποια παρανόηση. Δεν είπα ότι θα ήθελα να μεταρρυθμίσω την Όλαφ σε έναν οργανισμό. Είπα ότι ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει ανοιχτό πνεύμα για συζητήσεις, διότι ξέρω ότι διεξάγονται συζητήσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει αν δεν είσαι ανοιχτό, αν το πνεύμα ε, που έχει, που θα, ε, με το οποίο θα διέπει αυτέ τι ε, δραστηριότητε δεν θα είναι ανοιχτό, τότε δεν θα μπορεί να, είναι, να υπάρχει διαφάνεια. Και τώρα το να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα έχει προτερήματα για την Όλαφ. Είναι κοντά σε ένα μεγάλο θεσμικό όργανο, κοντά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να έχει προτερήματα αυτό. Έχει πρόσβαση κανείς σε όλα τα ε, στοιχεία και τις ε, έδρες και περιοχές εκτός ε, Ευρώπης. Έχει τη συνεργασία των Γενικών Διευθυντών και έχει στενή συνεργασία με την ITAC. Α, τώρα, από την άλλη πλευρά, και υπάρχει και το προτέρημα του να έχει κανείς πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία, στα, στις Αν δεν είναι κανείς τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε το πιο σημαντικό πρόβλημα θα μπορούσε να είναι ότι δεν θα είχε κανείς πρόσβαση άμεσα στις πληροφορίες, όπως έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες τώρα. Δεν εξέφρασα μια διαφορετική άποψη. Είπα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για τέτοιου είδους συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Αυτό ήταν όλο που είπα. Αυτό είναι αυτό το οποίο αναμένατε. Σας ικανοποιεί η απάντηση. Θα προσπαθήσω δύο ερωτήσεις σε ένα λεπτό να τις τριμώξω στη διατύπωσή τους είσαστε αστυνομικός υπάλληλος, έτσι δεν είναι αξιωματούχος αστυνομίας και υποθέτω ότι και στο σώμα αστυνομίας του Βελγίου υπάρχει και ένα τμήμα εσωτερικών εξεταστικών δραστηριοτήτων. Η Όλαφ είναι και ένα τμήμα εσωτερικών ακριβώς διακριβώσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Βέλγος αστυνόμος, αν σας πρότεινε κανείς εσωτερικές τέτοιες δραστηριότητες να εξαιρεθούν, πόσο πρόθυμος θα είσαστε για κάτι τέτοιο. Το δεύτερο, ακούσαμε έναν υποψήφιο που προέρχεται από την Όλαφ Ακούσαμε έναν υποψήφιο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα του ευρωπαϊκού παιχνιδιού ως ευρωβουλευτής παλαιότερα πολύ καλά. Ε, για σας τώρα θα ήθελα να μάθω κάτι για τις γνώσεις σας, τις δεξιότητες προσόντατας και τις ικανότητές σας σε σχέση με τα θεσμικά, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εργάζεστε με αυτά που είναι αρκετά περίπλοκα όπως θα γνωρίζετε ήδη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση, δεν έχουμε μία υπηρεσία, έχουμε δύο, που είναι πολύ καλή ιδέα θα έλεγα. Στην δική μου διεύθυνση και στην διεύθυνση εσωτερικών ερευνών, κάνουμε, ασχολούμαστε ακριβώ με αυτό. Δεν είναι καλή ιδέα το να υπάρχουν τρει διαφορετικέ ε, υπηρεσίε που ασχολούνται με εσωτερικέ έρευνε. Είναι καλή ιδέα το να υπάρχει μία υπηρεσία. Σε αυτό είμαι σαφής. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν αυτά από την ε, Όλαφ. Έχετε δίκιο. Δεν έχω την ίδια εμπειρία όπως οι άλλοι υποψήφοι που έχουν συνεργαστεί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για 10 χρόνια. Ε, τα τελευταία 10 χρόνια έχω μια συγκεκριμένη εντολή που αφορά το προσωπικό, τον προϋπολογισμό ή τους τομείς. Η διεύθυνση είναι παρεμφερή, η διεύθυνση μου παρεμφερής ε, με αυτή της Όλαφ. Λόγω αυτού, λόγω της συγγένειας ε, με την Όλαφ, υπήρξε σημείο επαφής για το Βέλγιο και για άλλες χώρες, για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου μου. Έχω λοιπόν πολλές επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή, με την Όλαφ, με πάρα πολλές γενικές διευθύνσεις. Έχω συναδέλφους που έρχονται στο ε, ε κοινοβούλιο Έχω συνεργαστεί με αυτούς τους συναδέλφους και σε αρκετές περιπτώσεις μου ζήτησαν να, να είμαι βασικός ομιλητής. Ήμουν λοιπόν ε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε όλους αυτούς τους τομείς. Πήρα μέρος στις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, κάτι που δεν ήταν εύκολο, αλλά με αυτόν τον τρόπο έκτισα μεγάλη πείρα. Έχω τη φήμη ανθρώπου που ξέρει να επιτυχάνει συμβιβασμούς. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να μην έχω την ίδια εμπειρία με τους υπόλοιπους υποψήφιους αλλά δίχως άλλο είμαι εμπειρος και το πλεονέκτημα είναι ότι έχω πολύ ανοιχτό μυαλό κάτι που είναι πλεονέκτημα γιατί νομίζω ότι μετά από 11 χρόνια είναι η ώρα να αλλάξουν τα πράγματα στην Όλαφ. Deutsch. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε πρόεδρε κύριε υποψήφιε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σκέψη αυτό το πρόγραμμα των 100 ημερών που θα υποβάλλεται. Με ένα νέο γενικό διευθυντή, όπως το γενικό διευθυντή Σόλαφ, αυτό είναι πολύ καλό. Μπορείτε να λογοδοτήσετε και με αυτόν τον τρόπο έναντι του προγράμματος αυτού. Μπορούμε να μετρήσουμε, να σταθμίσουμε το έργο που θα έχει επιτελεστεί. Σαν συνέπεια τούτου θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα αν και όταν εσείς γίνετε ο νέος ε, Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, αν μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα, πώς το βλέπετε, εσείς ε, θα δράσετε, θα μεριμνήσετε, ώστε οι κανόνες να αλλάξουν. Θα είναι αναγκαίο να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Οι διατάξεις, οι κανόνες, οι κανονισμοί θα πρέπει να αλλάξουν ή όχι. Διότι αυτές οι κανόνες και οι κανονισμοί θα μπορεί από πλευρά τη ίδια τη αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν λόγω αυτή τη επιθυμία του. Έχετε εσεί ε, σε σχέση με τον προπολογισμό τη όλα τον θεωρείτε επαρκή, θεωρείτε τα στελέχη που έχει Όλαφ αρκετά. Η πραγματογνωμοσύνη τη Όλαφ είναι επαρκή όσο έχει αυτή τη στιγμή. Πώς τα βλέπετε. Θα θέλατε να αναδομηθεί η Όλαφ. Θα θέλατε μεγάλες αλλαγές να γίνουν σε σχέση με τα στελέχη όσον αφορά τη δομή τους. Ευχαριστώ. Thank you very much for the question, sir. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που διαπιστώσατε ότι θα είμαι υπόλογος, διότι είμαι υπόλογος και στον τομέα μου. Έχουμε ε, πενταετές θητείες και ανανεώθηκε η θητεία μου και ε, θεωρήθηκα υπεύθυνος, ανανεώθηκε από την 1η Φεβρουαρίου. Λοιπόν, κατόπιν τούτου θέλω να σας πω ότι γνωρίζω πολύ καλά το πρόγραμμά μου είναι φιλόδοξο. Αλλά όχι επειδή είναι φιλόδοξο, θα πρέπει να αλλάξω τους κανονισμούς ώστε να πραγματοποιήσω το πρόγραμμά μου. Σε το χρόνο είμαι βέβαιος και γι' αυτό είπα ότι στο επιχειρησιακό μου σχέδιο έχω το βράχι μέσο και μακροπρόθεσμο. Σε το χρόνο κάποιοι κανονισμοί θα πρέπει ίσως να αλλάξουν. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά και χωρίς να αλλάξουμε τους κανονισμούς. Πάλι, ορισμένα παραδείγματα. Εάν θέλετε να επαναπροσδιορίσετε τις ε, διευθύνσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί. Αυτό είναι εσωτερικές διαδικασίες που μπορούν να γίνουν με την Επιπτική Επιτροπή. Μπορείτε να, να διευθετήσετε καταστάσεις χωρίς να αλλάξετε τα πάντα. Βεβαίως, το, τίθεται το θέμα του προπολογισμού. Από όσο βλέπω τώρα, δεν νομίζω μας χρειάζονται επιπλέον χρήματα στον προπολογισμό. Δεν μας χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Έχουμε αρκετά άτομα. Το θέμα είναι και αυτό είναι σύμφωνα με την εμπειρία μου. Το θέμα είναι έχουμε τα σωστά προφίλ. Εάν βλέπω ότι βλέποντας ότι υπάρχουν μόνο 35% του προσωπικού κάνει έρευνα και το 65% υποστηρικές εργασίες για μια ερευνητική μονάδα, αυτό είναι αδιανόητο. Θα πρέπει να αλλάξετε λίγο τη διάταξη, να, τα στοιχεία αυτά. 65% θα πρέπει, 65% θα πρέπει να ασχολούνται με έρευνα. Πρέπει λοιπόν να είναι πιο αποδοτικοί οι υπάλληλοι. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ξεχωριστή μονάδα για την προκαταρτική έρευνα, την αξιολόγηση των φακέλων, ώστε να υπάρχουν ειδικοί που θα κάνουν μόνο αυτό όλη την ημέρα, το οποίο σημαίνει ότι θα εξοικονομήσετε πόρους από άλλες μονάδες. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε αρκετά χρήματα, αρκετό προσωπικό και αρκετή εμπειρία. Ναι, θα πρέπει πρέπει να αναδιαρθρωθεί η ΟΛΑΦ, διότι προς το παρόν, ως έχει σήμερα, η ΟΛΑΦ δεν έχει σωστή διάρθρωση με το σωστό της αντικείμενο που είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαίων και η διεξαγωγή ερευνών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμα υποψήφια στην παρουσίασή σας είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί καλή συνεργασία, θετική συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή, καθώς βρίσκεται η μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση καθοδών, διαρκώς κάνουμε λόγο για την ανάγκη να είναι πιο στενή η συνεργασία με τα υπεύθυνα αρμόδια θεσμικά οργάνα των κρατών μελών. Υπάρχει και μια πρόταση να ενταχθεί στον κανονισμό, να συμπεριληφθεί ότι τα αρμόδια θεσμικά όργανα των κρατών μελών θα πρέπει να ενημερώνουν την Όλαφ για περιπτώσεις ε, έρευνας ε, μία φορά ε, αναέτος ή μία φορά αναεξάμεινο ή όταν αυτό θα είναι αναγκαίο σε σχέση με την Όλαφ. Ποια είναι η δική σας άποψη, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία για να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διακριβωτικές εργασίες στο μέλλον και για να αποφύγουμε του να έχουμε περιορισμένες ε, διοικητικές τέτοιες δράσεις ε, που δεν θα είναι αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για, τις ερωτήσεις, για την ερώτησή σας κύριε. Θα έλεγα από πλευρά μου ότι η καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι ένα σημείο που έχει σημασία κλειδιού για το μέλλον της ε, όλα Πολλές από τις δραστηριότητες σήμερα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες επειδή η Όλαφ εργάζεται υπερβολικά μεγάλο διάστημα επ' αυτών. Έχω παρακολουθήσει το θέμα. Όταν έρχονται στο Βέλγιο πολύ συχνά δεν υπάρχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αυτές τις εξεταστικές δραστηριότητες διότι επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν εξεταστεί αυτά τα θέματα και το ενδιαφέρον έχει πλέον απολεστεί. Εγώ θα ήμουν υπέρ μεγαλύτερη στενότερης συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και ταχύτερης ανταλλαγής πληροφοριών. Έχουμε την δυνατότητα τώρα να έχουμε μια κοινή εξεταστική τέτοια δραστηριότητα. Το έχουμε κάνει αυτό και ήταν πολύ επιτυχές στο παρελθόν. Σίγουρα λοιπόν αυτού του είδους ε, η προσέγγιση ιδιαίτερα όταν ε, αφορά αυτό την Όλαφ είναι, έχει τεράστια σημασία και γι' αυτό και πάλι τώρα πρέπει να ανασχεδιαστεί η ε, λειτουργία της α, Όλαφ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στενοποί και υπάρχουν δυσκολίες για να ολοκληρωθεί μια δραστηριότητα και θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Χρειάζεται και εδώ θάρρος σίγουρα το έκανα αυτό στη γενική μου διεύθυνση πριν από 10 χρόνια όταν ήμουν ε, γενικός διευθυντής. Ε, ήμουν νεότερος τότε. Δεν θα ήταν δυνατόν να το έκανα τώρα. Αν το έκανα τώρα το ίδιο το δικό μου δημιούργημα ε, θα το οδηγούσα σε αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτό σε σχέση με την Όλαφ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για το θάρρος σας Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερη τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας υψηλός αξιωματούχος από την αστυνομία να θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εργαστεί για αυτήν. Μας τιμά αυτό. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θάρρος το οποίο έχετε. Όταν λέτε ότι 35% είναι ερευνητικές δραστηριότητες και είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες οι περιπτώσεις και αυτό καλό το οποίο είπατε. Παρόλα αυτά έρχεστε από την αστυνομική υπηρεσία. Ο, ο Όλαφ είναι ένα θα έλεγα ερμαφρόδιτο δημιούργημα. Είναι ένα ξεχωριστό δημιούργημα. Πόσο πολιτικά εμπνέεστε εσείς, πόσο πολιτικός είναι ο ρόλος της Όλαφ σύμφωνα με την άποψή σας. Διότι δεν είναι μόνο εξεταστικέ οι δραστηριότητες εσείς, έχει και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Παρότι εδώ ίσως υπάρχει υπερβολική θα έλεγα επικέντρωση σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω από πλευράς της πείρας μου στην γενική μου διεύθυνση. Έχουμε διαφορετικές ε, ε, ε, ομάδες, ενότητες. Είχαμε στην την, υψη, την Ανώτατη Επιτροπή Εποπτείας που είχε ακριβώς την ίδια δομή όπως έχει η όλα τώρα, διοικητικές λειτουργίες. Δεν ήταν αστυνομική δύναμη, ήταν ε, πολύ κοντά πάλι και αυτό, αυτή η μονάδα, αυτή ε, η ε, δομή στην πολιτική στάθμιση των πραγμάτων. Έχω λοιπόν την πείρα πώς μπορεί μια αστυνομική, μια τέτοια δύναμη να μεταμορφωθεί. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον μέλλον, ποιο θα είναι το μέλλον, ποιο θα είναι ο ρόλο στο μέλλον τη Όλαφ. Το πιο σημαντικό θέμα είναι σε σχέση με την, δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι πιθανότατα, πιθανότατο να μπορέσει να συνεργαστεί η Όλαφ ως τμήμα αυτής της εισαγγελίας με τη Europol και την Eurojust. Η Europol θα συλλέγει τις πληροφορίες και τα στοιχεία και η Eurojust θα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ας το πω έτσι, το τμήμα ε, το δικαστικό. Αυτό σίγουρα θα έχει σαν συνέπεια ότι η επιρροή των πολιτικών Τη της πολιτικής στην Όλαφα θα μειωθεί. Όμως στο μεσοδιάστημα φυσικά πρέπει να ζήσουμε με την ίδια την πραγματικότητα, να την δεχτούμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό από πλευρά του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Όλαφ το ίδιο ακριβώς όπως κάνω στη γενική μου διεύθυνση εγώ τώρα. Δεν επιτρέπω με κανένα τρόπο η πολιτική να αναμειγνύεται στις δραστηριότητές μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και κάνω λόγο εδώ για την πολιτική ανάμειξη στις δραστηριότητές μας. Όταν κάνουμε λόγο για την πολιτική, την πολιτική ζωή, το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν το δικό τους ρόλο και πρέπει να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τις απόψεις τους και να προσπαθούμε να βρούμε τις σωστότερες λύσεις. Όσον αφορά δραστηριότητες και τις εξετάσει εξεταστικές δραστηριότητες η όλα αυτά πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητοι χωρίς πολιτική ανάμειξη. Ο κύριος Στάις παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς κύριε έχετε μακρά πείρα στο Βέλγιο και έχετε και πολύ καλή φήμη και έχετε και προτερήματα και τα αναφέρατε αυτό ότι μέσα στο πλαίσιο του έργου σας εσείς με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με την Όλαφ είχατε στενή επαφή και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον όπως το ανέφεραν και άλλοι υποψήφοι ήταν ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από εσά. θέσατε το κέντρο βάρους στις πραγματικές εξεταστικές δραστηριότητες είπατε από το 35% δεν επαρκεί αυτό πρέπει να υπάρξει αύξηση να υπάρξει μετά διάθεση σε 50%. Αυτό αφορά όμως ε, και συγκεκριμένες δραστηριότητες τη Όλαφ που θα πρέπει με διαφορετικό τρόπο να ασκηθούν. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, να μας εξηγήσετε περισσότερο αυτές τις απόψεις σα Το ίδιο ακριβώς ε, ισχύει και θα πρέπει κανείς το βάρος των περιπτώσεων να το δει κανείς. Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα θα ήθελα να πω, έχω κάτι παρόμοιο, κάτι παράλληλο, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Η de πολιτική της Όλαφ είναι ένα πολύ καλό μέσο. Μπορεί κανείς να έχει κατόφλια για το τι κάνει και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται κάποιες υποθέσεις. Και από εκεί μπορεί κανείς να δει αν ναι ή όχι κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να τύχουν συνέχεια και εξεταστική ε, δραστηριότητα περαιτέρω. Το ίδιο και σε σχέση με τις εσωτερικές ε, διακριβώσει. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον από τα κράτη-μέλη μπορεί να διαπραγματευτεί, να διαβουλευτεί κανεί με τα κράτη-μέλη και να ε, δει κανεί σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες τι πρέπει να γίνει. Μπορεί να υπάρξει συσσόρευση τέτοιων ε, περιπτώσεων ή μπορεί να υπάρξει μετάθεση τέτοιων περιπτώσεων στα κράτη-μέλη ώστε να απελευθερωθούν ε, κονδύλια και στελεχειακό δυναμικό για άλλες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξουν περισσότερες, περισσότερες επενδύσεις στις, δραστηριότητε εξεταστικές δραστηριότητες και να τεθούν προτεραιότητες ιεραρχώντας για την Όλαφ. Το χαρτοφυλάκιο αυτή τη στιγμή των δραστηριοτήτων είναι υπερφορτωμένο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να περάσει κανείς ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο με την τεμήνιμης πολιτική που δεν θα μπορούσε να έχει τις ίδιες προδιαγραφές για τους ε, διαφορετικούς τομείς ε, με τους οποίους ασχολείται η Όλαφ σήμερα. Θα ήταν διαφορετική προσέγγιση για τα διαθωτικά ταμεία σε σχέση με τα τελωνία, για παράδειγμα. Όμως οι ίδιοι κανόνες και κανονισμοί για τους διαφορετικούς τομείς πρέπει να εφαρμόζονται. Αν το κάνει κανείς αυτό και έχει αυτή τη διαφοροποίηση θα μπορέσει να μειώσει το βάρος, τον όγκο των περιπτώσεων. Και κινώντας από αυτό το σημείο είναι σημαντικό, θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα στρατηγικό για το πώς θα μπορεί να δοθεί συνέχεια σε αυτά. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία σε σχέση με τους επικεφαλείς μονάδων και τομέων. Τρίτον, θα πρέπει πολύ πιο γοργά να εμπλέκεται η δικαστική αρχή, η, ε, ε, οι διοκτικές αρχές να μπορούν να εμπλέκονται ώστε να μην ακολουθηθεί η λανθασμένη τροχία. Και στο τέλος τέλος είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μετάθεση νωρίς σε πρώιμη φάση στα κράτη-μέλη και μπορεί και κοινή ομάδα, ε, εξεταστική ομάδα να δραστηριοποιηθεί Όλαφ και κρατών μελών. Και αυτό θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει και θα μπορέσει έτσι να ανακτηθούν, θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε ε, πόρου και κονδύλια και είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί με του οποίου μπορούμε να μειώσουμε το βάρο ε, των περιπτώσεων αυτών, του αριθμού των περιπτώσεων. Νομίζω δεν είναι κανεί από την ομάδα ΙΣΙΑΡ, συνάδελφο Σερενάουζερ. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάντα, όχι όμως πάντα, καμιά φορά υπάρχουν κάποιες διαφορετικές περιπτώσεις. Καμιά φορά έχουμε ε, περιπτώσεις και στοιχεία τα οποία δίνονται στα μέσα του τύπου, ε, στα μέσα ενημέρωσης και έτσι παραβιάζονται κάποιες αρχές. Από την άλλη πλευρά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπάρχει απουσία διαφάνειας καμιά φορά. Θα λέγατε ότι αυτά είναι οξυμένα προβλήματα τα οποία εσείς ως Γενικός Διευθυντής θα θέλατε να αντιμετωπίσετε και με ποιες αρχές με ποια ε, προσέγγιση θα αντιμετωπίζατε την αρχή της εμπιστευτικότητας ε, αναπερίπτωση θα την αντιμετωπίζατε ή θα είχατε ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης μια ενιαία αρχή που θα σας διείπε στη δράση σας. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι ένα πρόβλημα και πρέπει να έχεις μια πολιτική σε ένα θεσμό, πρέπει να υπάρχει εταιρική πολιτική. Στη δική μου τη διεύθυνση το ίδιο συμβαίνει. Ε, υπάρχει η χεμήθεια, η χεμήθεια και το απόρριτο είναι πολύ σημαντικά. Βεβαίω η διαφάνεια χρειάζεται, αλλά πρέπει να τη δώσετε το σωστό χρόνο ενώ σου εξελίσσεται μια υπόθεση δεν μπορεί να κοινοποιηθεί τίποτα στον τύπο από τα άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτή την έρευνα. Στο τέλος πρέπει να εξασφαλίσετε τη διαφάνεια στο τέλος έρευνας και το σημαντικό είναι να δείτε ποιον θα φυλάξετε ως εποπτικό όργανο η Όλαφ πρέπει να το γνωρίζει να διασφανίζει δηλαδή το απόρριτο και τη διαφάνεια πιστεύω λοιπόν ότι τα δικαιώματα των ατόμων που βρίσκονται υπό έρευνα είναι πολύ σημαντικά και το, τα δικαιώματα των πληροφοριοδοτών. Από την αρχή λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια ώστε να διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων Υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η Υποπτική Επιτροπή. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο τη Υποπτική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι πολύ καλή άσκηση γίνεται εδώ, πολύ καλή δουλειά γίνεται από το Κοινοβούλιο, διότι μπορεί κανείς να κάνει μια καταγγελία για θέματα διαδικαστικά. Ε, ε, έτσι υπάρχει μια εγγύηση για την ορθότητα τη σωστή διενέργεια ε, της έρευνας για την εχεμήθεια της έρευνας και μπορείτε συγχρόνως όμως να επιδείξετε απόλυτη διαφάνεια αλλά τη σωστή στιγμή στο πέρα της έρευνας τη στιγμή που έχει μεταφερθεί πλέον στο πλαίσιο των κρατών μελών, τα οποία θα αποφασίσουν για το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι μια γενική πολιτική που θα ακολουθούμε. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. 36 μήνες ε, κατά μέσον όρο, τρία χρόνια δηλαδή διαρκεί, μέχρι ότου αναφερθούν τα κράτη-μέλη για περιπτώσεις ε, παρατυπιών στην Όλαφ. Είσαστε από το Βέλγιο και το Βέλγιο είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος ε, της λύσης. Υπάρχει μικρή προθυμία της δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην Όλαφ για την εξέταση περιπτώσεων. Εμείς ως Κοινοβούλιο υποβάλαμε κάποιες μεταρρυθμιστικές προτάσεις. Θα με ενδιαφέρει να ξέρω με αυτές τις προτάσεις μπορούμε να βασιστούμε στη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ. Uh, uh, Να απαντήσω πρώτα όσον αφορά το θέμα του Βελγίου. Επειδή βρίσκομαι πολύ κοντά ε, στην εισαγγελία του Βελγίου και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα, το πρόβλημα είναι το εξή. Επειδή η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο Βέλγιο, περίπου τα, οι μισές περιπτώσεις ε, καταλήγουν στη βελγική δικαιοσύνη. Και εδώ έχουμε πρόβλημα πόρων και συχνά καταφθάνουν στη δική μου τη διεύθυνση. Και σας εγγυώμαι ότι αν ε, η εισαγγελία τα δέχεται, δέχεται αυτές τις υποθέσεις, διότι μπορούν να αποφασίσουν να μην τις δεχθούν, εγώ πάντοτε δίνω προτεραιότητα σε αυτές τις υποθέσεις, τις όλα δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό έχει καλό αποτέλεσμα. Το δεύτερο σκέλος ερώτησής σας τώρα. Ότι το Κοινοβούλιο έκανε μια σχετική πρόταση. Οι προτάσεις του Κοινοβουλίου είναι πολύ καλές, πιστεύω, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, αναφέρεται στην πρόταση του, της ε, ε, προσαρμογής του, των κανόνων του 1999 και λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα της υπεράσπισης πολύ σωστά και των πληροφοριοδοτών Επίσης, ε, διευκρινίζεται ποιες είναι οι εγγυήσει όσον αφορά τη διαδικασία. Θέλετε να έχετε πιο αυστηρούς κανόνες έρευνας, να καθορίσετε με σαφήνεια το ρόλο της Εποπτικής Επιτροπής, που είναι κάτι το απαραίτητο μετά από 11 χρόνια διότι αυτό θα φέρει την ΟΛΑΦ στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και είμαι πολύ ευτυχής με τις προτάσεις σας και νομίζω η καλύτερη πλευρά είναι το θέμα ε, του να υπάρχει ένα σύμβουλος που θα προστατεύει τις διαδικασίες τις οποίες θέλει να προσαρμόσει όλα. Υπάρχει μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Αναφερθήκατε σε ένα πρόγραμμα ευρείας κλίμακας. Η ερώτηση μου είναι ποιος είναι ο πρώτος τομέας που θα ευνοηθεί από αυτή την επέκταση. Συγγνώμη, δεν έφτασε η μετάφραση, δεν κατάλαβα την, ε, το πρώτο. Αναφέρουμε στο πρόγραμμα Πλούτο. Ωραία, το πρόγραμμα Πλούτων. Το ξέρω το πρόγραμμα Πλούτων και ξέρω ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα στον τομέα της ε, πρόληψης. Θα, μπορούσαμε, θα μπορούσε να ενισχύσει τις ε, προσπάθειές μας ακόμα περισσότερο για να καταπολεμήσουμε την απάτη. Βεβαίως υπάρχουν τομείς που θα εκμεταλλευτούν αυτό. Μιλώντας ε, για συνεργασία πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών από τις χώρες μέλη. Οι χώρες μέλη έχουν τα, συγκεκριμένους τομείς ε, που έχουν συμφέροντα, για παράδειγμα γεωργία ή τελωνία. Όπου υπάρχουν συμφέροντα δίνουν εύκολα πληροφορίες. Υπάρχουν όμως και άλλοι τομείς που δεν τους ενδιαφέρουν και δυσκολεύονται να δώσουν πληροφορίες. Εκεί ακριβώς θα μπορούσε ο Πλούτον να παίξει σημαντικό ρόλο. Εάν θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα δίχως άλλα τα αποτελέσματα θα ήταν πάρα πολύ καλά. Ανδρέας. Κύριε Ανδρέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντενόλφα, τονίσατε τις, ικανότητες, τις πολιτικές και διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Ο συνάδελφος ε, κύριος Χατζημαρκάκης έθεσε μία ερώτηση για τις πολιτικές σας δεξιότητες. Η η προστασία των οικονομικών συμφερόντων δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Σε τι βαθμό θεωρείτε αυτές τις πολιτικές και οικονομικές ικανότητες σημαντικές για το ρόλο αυτό του Διευθυντή της Όλαφ. Δεύτερον, Συγγνώμη, θεωρείτε ότι οι εσωτερικοί πληροφοριοδότες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο έργο σας. Ιδιαίτερα ικανοποιημένο είμαι που διατυπώνετε αυτή την ερώτηση. Τώρα, σε σχέση με τι ε, πολιτικέ μου ικανότητε, ε, έχω τη φήμη ότι είμαι καλό διαχειριστή ε, και ότι είμαι ισχυρό όσον αφορά τα θέματα τη πολιτική στοχοθέτηση. Όμως ειλικρινά έχω ελευθερία δράση σε σχέση με την πολιτική πτυχή. Δεν υπάρχει κάποια, α το πω έτσι, μεροληψία σε σχέση με κάποιο πολιτικό κόμμα Ίσως υπάρχει κάποια παρανόηση λοιπόν εδώ. Τώρα, σε σχέση με την ε, δική μου, ας το πω έτσι, τα δικά μου χαρακτηριστικά, έχω ιδιαίτερα ισχυρά χαρακτηριστικά διαχειριστή και έχω και φήμη καλού διαχειριστή. Και έχω την, ε, ε, ας το πω έτσι, φήμη ότι μπορώ να διαπραγματευτώ με πολιτικούς για να πετύχω αυτό το οποίο θέλω είναι διαφορετικό αυτό από εκείνο το οποίο εσείς ε, εννοούσατε. Νομίζω θα έπρεπε να έρθω σε αυτό το θεσμικό όργανο και να διαπραγματευτώ και να συζητήσω. Θα πρέπει να είμαι ανοιχτό και διαφανής ε, για τη σκέψη σας και τον τρόπο του σκέπτεστε το δικό σας. Αυτή είναι η δική μου ε, πρώτη τοποθέτηση. Και όσον αφορά την αξιολόγησή μου για τους πληροφοριοδότες εκ των έσω, φυσικά είναι σημαντική αυτή και υπάρχουν κανονισμοί και από πλευρά προσωπικού για την, τα, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δύο άρθρα κανονισμού για τους εσωτερικούς πληροφοριοδότες. Ένα πράγμα λείπει όμως. Δεν υπάρχει τίποτα όμως που να προστατεύει αυτούς τους πληροφοριοδότες υστερότερα. Και αυτό είναι σημαντικό όμως. Πρέπει να υπάρχει προστασία όμω δεν προβλέπεται κάποια τέτοια προστασία. Είναι σημαντικό όμω το θέμα τη προστασία και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπένοφ. Καλό σας βράδυ. Ας ακούσουμε τώρα την τέταρτη υποψήφια, την κυρία Κριστίνα Γκέλερμπραντ, που θα θέλαμε να χαιρετήσουμε και θα ήθελα να της δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Κυρία Γκέλερμπραντ. Good afternoon. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιαστώ σε εσά και να σας πω τις απόψεις μου για την Όλαφ. Ονομάζομαι Κριστίνα Γκέλεμπραν Χάγκμπεργκ. Είμαι δημόσιο υπάλληλο, αφοσιωμένο από, από το κράτος μέλος Σουηδία και έχω τη φιλοδοξία να γίνω επικεφαλής ε, της ΟΛΑΦ. Λοιπόν, ξεκινάω με τα γεγονότα. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέα ούτε δικαστή. Δεν έχω επαγγελματική εμπειρία από εργασία στι Βρυξέλλε και δεν έχω εργαστεί στα πλαίσια τη ΟΛΑΦ. Αλλά είμαι Υπαριθμόν ένα, ικανή outsider, έχω μάστερ νομικής, με σημαντικές διοικητικές και πρακτικές εμπειρίες, με θάρρος να σταθώ ακόμα και όταν ο άνεμος γίνεται θύλα, με ένα όραμα να αναλάβω μία από τις πιο δύσκολες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω επιτυχημένη καριέρα στην καταπολέμηση και την πρόληψη της διεθνούς απάτης σε μια οργάνωση παρόμοια με την Όλαφ, διπλάσια όμως από την Όλαφ και με διπλάσιο προπολογισμό και πάντως σε συνεργασία με, τα κράτη, με συναδέλφους από τα άλλα κράτη-μέλη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα παρακολουθώ, θα ενισχύω το διάλογο, θα εργάζομαι στενά με όλους τους ενδιαφερόμενους, αλλά θα ενεργώ ανεξάρτητα, διότι είμαι ένα ανεξάρτητο άτομο. Και θεωρώ την εξαρτησία της Όλαφ ως ουσιαστικό θέμα σε όλες τις έρευνες. Οι βασικές μου προτεραιότητες είναι οι εξής. Να υπάρξει σημαντική βελτίωση ποιοτική και σε αποτελεσματικότητα στις έρευνες και στις εργασίες της ΟΛΑΦ. Γι' αυτό θα εστιαστώ στη βελτίωση της ποιότητας της αποτελεσματικότητας φροντίζοντας ότι θα προστατεύουμε με προσοχή τα δικαιώματα όλων των ατόμων χρησιμοποιώντας τις άριστες πρακτικές και των μεθόδων εργασίας με ανάλυση κινδύνων και σωστή στρατηγική ελέγχου. Θα φροντίσω ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών θα συνοψίζονται, θα αναλύονται και θα αξιοποιούνται για όλου, ώστε να αποτρέπεται η απάτη και να προστατευόμαστε από την απάτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα εξασφαλίσω διαφάνεια και διάλογο με του ενδιαφερόμενους και με τις ε, οργανώσει αδελφέ όλο τον κόσμο, ώστε να αξιοποιηθεί η δύναμη τη ΟΛΑΦ για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όπω και με τον κόσμο γύρω μας, η Όλαφ θα πρέπει συνεχώ να αλλάζει για να αναπτύσσεται, να ανταποκρίνεται στι απαιτήσει του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντο και στι αυξανόμενε απαιτήσει και προσδοκίε για να αντιμετωπίσει επιτυχώ τη διαφθορά και την απάτη. Θα το επιτύχω με την εμπειρία μου και τι διαχειριστικέ μου ικανότητε, υποστηρίζοντα την κατάρτιση και την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών, για να βελτιωθούν οι επαγγελματικέ ικανότητε και τα κίνητρα που θα έχουν όλα τα άτομα μέσα στην Όλαφ. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για μια επιτυχημένη ιστορία. Είναι η ιστορία της Χαβάλα. Ένας τρόπος γρήγορος και αποτελεσματικός για να αποστέλλονται χρήματα, για να μεταφέρονται χρήματα και εκτός του συστήματος της κοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση φρόνησα ώστε οι πόροι πολλών ε, αρχών να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά ανακαλύπτοντας ότι το σύστημα μεταφοράς χρημάτων χρησιμοποιείται για, εγκληματικέ για εγκληματικές δραστηριότητες. Γι' αυτό πολλές χαβάλες ερευνήθηκαν και χρησιμοποίησα την, ε, τις πληροφορίες βασιζόμενοι σε στοιχεία όπως ε, εκθέσεις από τράπεζες ή από άλλα ιδρύματα μεταφοράς χρημάτων. Σε μια περίπτωση διαπίστωσα ότι μια εταιρεία η οποία οργάνωσε μεταφορές χρημάτων από τη Σουηδία υπάρχουν πολλοί τρόποι να μεταφέρει κανείς χρήματα ένομα από αυτή τη χώρα. Το διαπίστωσα λοιπόν, επειδή η εταιρεία δεν πλήρωνε φόρους και επίσης στα λογιστικά τους βιβλία δεν τηρούσαν τους κανόνες των διεθνών συναλλαγών. Είδαμε ότι χιλιάδες συναλλαγές, 120 εκατομμύριων ευρώ, σε 25 διαφορετικούς λογαριασμούς, σε τέσσερις μεγάλες τράπεζες, ε, δεν ήταν σωστές και κατασχέθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ιδιοκτήτη εταιρεία τιμωρήθηκε ε, για τέσσερα χρόνια, με τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Εάν μου δώσετε την εμπιστοσύνη και γίνω η επόμενη Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, σκοπός μου είναι να γίνει επικεφαλής οργάνωση σε όλο τον κόσμο για την καταπολέμηση απάτης. Και δεν σα υπενθυμίσω ότι όταν αποφασίσετε για τον επόμενο Γενικό Διευθυντή να έχετε υπόψη σας ότι ο, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές όπω ο Μαραντόνα δεν σημαίνει ότι είναι και οι καλύτεροι προπολιτέ. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Μη σα ευχαριστούμε, κυρία Γκρέσ, παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δυναμική γυναίκα. Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη ματιά. Έχετε δίκιο με το θέμα του προπονητή και του ποδοσφαιριστή. Βεβαίως ισχύει και το αντίθετο. Εσείς σε κάθε περίπτωση είστε ειδικοί σε θέματα οικονομικά και προέρχεστε από μια χώρα που πραγματικά έδωσαν αγώνα κατά της απάτης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι αλλαγές που σκοπεύετε να προωθήσετε στην Όλαφ εδώ και 11 μήνες ε, δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνο, κάποια διεύθυνση. Ποια κατά την άποψή σας είναι τα σημαντικά μέτρα. Okay. Uh, I believe that I don't... Ενδεχομένως δεν είναι συνήθιτα τα χαρακτηριστικά μου ή τα προσόντα μου για αυτή τη θέση. Κοίταξτε όμως, έχω σπουδάσει νομικά, μολονότι δεν εργάστηκα ποτέ σε ένα δικαστήριο. Κατά την άποψή μου, και αυτό με βάση τις πληροφορίες που έχω από την Όλαφ, τι αιτήσιε εκθέσεις αλλά και ορισμένες επικρίσεις που διάβασα στον τύπο, πιστεύω ότι όλα χρειάζεται έναν διαχειριστή που θα μπορέσει να επιφέρει αλλαγές στην οργάνωση. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε όχι για νομικές ικανότητες, αλλά για διαχειριστικές ικανότητες. Οι αλλαγές θα γίνουν, πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο για την Όλαφ. το μελέτησα το πλαίσιο και διαπίστωσα ότι το υπάρχον πλαίσιο δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Όπως είπατε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβράδυνε την πορεία της Ιόλαβ και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι. Ήμουν υπέρ μεγάλων οργανώσεων και εκεί κατάφερα να τις βοηθήσω να προχωρήσουν και νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω και την ε, Όλαβ. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία και να δούμε τι ακριβώς απαιτείται. Μία οργάνωση που έχει το μέγεθος της Όλαβ απαιτεί και μία ομάδα που θα είναι ικανή για να επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Αυτό μπορεί να γίνει και ορισμένες από αυτές τις αλλαγές μπορούν να γίνουν άμεσα. Το η δική μου πρόταση είναι το να γίνει ένα πρόγραμμα τριετές και πενταετές. Έχουμε ένα αξίωμα στην Όλαφ που διαφορετική στοχοθέτηση πρέπει να ακολουθεί. Εσωτερικές έρευνες, εξωτερικές έρευνες, ασχολείται με μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, κατά των απατών με κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς ε, των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πιθανώς αυτά τα συμφέροντα θίγονται. Ερώτησή μου, πώς βλέπετε την ισορροπία αυτών των διαφορετικών τομέων στους οποίους εργάζεται η Όλαφ βλέπετε να υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές ή αναδιαρθρώσεις. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι αλλαγέ είναι αναγκαίε παντού. Σήμερα η όλα δαπανά το 12% των πόρων για εσωτερικέ έρευνε. Ενδεχομένω αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να τα δω από κοντά τα πράγματα, να μιλήσω για αυτού που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση. Όπω γνωρίζετε, είμαι δημόσιο υπάλληλο εργάστηκα στον, ε, σε, φορο, σε φορολογικές υπηρεσίες. Τα τελευταία δέκα χρόνια συνεργάστηκα με την αστυνομία σε εθνικό επίπεδο στην Σουηδία, αλλά για θέματα διακρατικά. Η πείρα με έχει μάθει το πώς να αντιμετωπίζω τα θέματα σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και μέσα στην Όλαφα. Να δούμε δηλαδή ποιοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και πώς θα συνεργαστούμε μαζί τους. Μία από τις βασικές αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν θα ήταν σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Φιέλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή η γλώσσα μας, να μιλήσω στα σουηδικά και θα το κάνω. Έχουμε συζητήσει λοιπόν πολύ για αυτά. Έχουμε συζητήσει για το ποιες αρμοδιότητες ακριβώς αξιολογούμε ιδιαίτερα μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχουν τρία πράγματα που για μένα έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Φυσικά πρέπει να είναι το κατάλληλο άτομο γενικά. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα προσόντα και ικανότητες αφενός πήρα όσον αφορά θέματα διαχείρισης. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο θα έλεγα και είναι πρόδειλο, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το αποδείξει κανείς. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα αρμοδιότητες και γνώσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα συνεργασίας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη δικαιοσύνη και τα δικαστικά. Θα ήθελα κάπως περισσότερο να μας λέγατε περισσότερα σε σχέση με αυτή την ευρωπαϊκή συνεργασία και σε σχέση και με τις δικαστικές έρευνες. Ευχαριστώ. You asked about the three areas. Αναφερθήκατε στους τρεις τομείς. Επειδή πρόσφατα μίλησα για την ε, διαχειριστικές μου ικανότητες, ας επικεντρωθούμε στις άλλους, στους δύο τομείς. Όχι, δεν έχω έργα στις Βρυξέλλες Ήμουν από την άλλη πλευρά. Εργάστηκα σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μου και ήμουν υπεύθυνη της ε, Εθνικής Αρμόδιας Αρχής. Αρκετά από τα μέλη του προσωπικού εργάζονται στον τομέα των ερευνών που έχουν ξεκινήσει από την Όλαβ. Αυτή, αυτό είναι ένας από τους τομείς που είμαι έμπειρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νομικές μου γνώσεις, Ασχολούμαι βασικά με το θέμα των φόρων. Επειδή όμως τα τελευταία 15 χρόνια ε, ήμουν σε υψηλόβαθες με θέσεις, είχα την δυνατότητα να εξετάσω διάφορους νομικούς τομείς και όπως είδατε από την, το βιογραφικό μου καθε 2 2-3 χρόνια άλλαζα θέση. Αυτό σημαίνει ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθώ είναι να εξοικειωθώ και με άλλους τομείς, μιλώντας πάντοτε για νομικά θέματα. Μπάστε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμη υποψήφια. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το θάρρος σας την γενναιότητά σας υποβάλλοντας ε, την υποψηφιότητά σας. Καθώς άκουσα η πείρα σας, η εμπειρία σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό έχουμε και, εδώ έχουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε έναν καλό προπονητή Μωρίνιο που αποδεικνύει ότι μπορεί κανείς να, να είναι καλός διαχειριστής και καλός προπονητής για παράδειγμα. Όσον αφορά το μέλλον και τις ε, αρχές που θα σας διέπουν στο έργο αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πολύ στενούς δεσμούς και συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη η Όλαφ. Σε ποιους τομείς πιστεύετε εσείς ε, ότι αυτοί οι δεσμοί θα πρέπει να βελτιωθούν και να συσφιχθούν περισσότερο σήμερα και στο μέλλον, διότι αυτό θα αναβαθμίσει την ποιότητα του, ε, της εργασίας της Όλαφ. Νομίζω ότι θα έξερε ένα σημαντικό θέμα για την όλα, στο μέλλον. Ένα από τα θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την Όλαφ είναι σε κάθε τομέα η Όλαφ θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με τη χώρα μέλος πολύ νωρίτερα από ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα. Όταν διαβάζουμε για τα αποτελέσματα στην Όλαφ, μερικές φορές Συνειδητοποιούμε ότι έχει περάσει πολλή χρόνο από τη στιγμή που ξένης ξεκίνησε η Όλαφ την έρευνα μέχρι τη στιγμή που ε, επιδόθηκε η έκθεση στη χώρα μέλος. Εάν ε, το διάστημα αυτό είναι δύο ετών, εγώ καταλαβαίνω τον ε, ανακριτή στη χώρα μέλος που θεωρεί ότι δεν θέλει να ξεκινήσει μια νέα περίπτωση γιατί βασιζόμενο σε παλιά δεδομένα. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα στο μέλλον είναι να ξεκινήσει συνεργασία με τις χώρες μέλη πολύ νωρίτερα, σε μια πολύ πιο πρώιμη ε, φάση. Ο κύριος Χατζημερκάκη. Κύριο Σμιτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Ξέρετε ότι εδώ κορεδεύουν και λίγο. Θα ήθελα να προσθέσω ένα επιπλέον κριτήριο εδώ. Η, στην Ευρώπη χρειαζόμαστε δυναμικές γυναίκες, πολλές δυναμικές γυναίκες. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα ορίσετε την ανεξαρτησία σε σχέση με την Όλαφ και το ρόλο της Όλαφ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έχουν τα πράγματα, η ανεξαρτησία έχει ως εξής. Η Όλαφ αποτελεί μέρος της Επιτροπής. Είναι μία οργάνωση η οποία ασχολείται με διοικητικές έρευνες ως υπηρεσία. Δημιουργήθηκε σε ένα... Ε, έχει αποφασιστεί σε νομικό πλαίσιο ο Διευθυντής της Όλαφ ως άτομο είναι ανεξάρτητος και οι έρευνες που γίνονται από την Όλαφ είναι ανεξάρτητες έρευνες. Για να υπάρξει μια εγγύηση της ανεξαρτησίας δημιουργήθηκε μια εποπτική επιτροπή. Τώρα, το κατά πόσον αυτό είναι παρκές για το μέλλον δεν μπορώ να το πω. Αλλά αυτό είναι το νομικό πλαίσιο που με απασχόλησε όταν ε, υπέβρα την υποψηφιότητά μου για τη θέση αυτή και έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Το, το, αν το όταν το κοινοβούλιο κάνει, υποδείξει κάτι, η όλα θα πρέπει να κινητοποιηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα γενικού διευθυντή της Όλαφ, αλλά εάν γίνει πρόταση για μία αλλαγή, δίχως άλλο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Στάς, κυρία υποψήφια, αναφέρατε το ποδόσφαιρο. Πολλοί ανταποκρίθηκαν και το κάνουν δύσκολο τώρα για μένα. Και εγώ από το Βέλγιο είμαι και σε σχέση με το ποδόσφαιρο δεν έχουμε τίποτα να επιδείξουμε. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν στο ποδόσφαιρο, δεν θα δώσω συνέχεια σε αυτό. Έχουμε έξι υποψηφίους από την άλλη πλευρά. Υποψηφίου για το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή τη Όλαφ. Τρεις... Ε, ε, από πλευράς ε, εσωτερικών δραστηριοτήτων έχουμε τρεις οι οποίοι είναι νέοι κατά το μάλλον ή σε σχέση με τις δραστηριότητες ε, αυτού του οργάνου που πρέπει να αποκτήσει περισσότερο οξυγόνο και να αναζωογονηθεί. Ασκήθηκαν επικρίσεις ε, και ακούστηκαν επικρίσεις σε σχέση με την Όλαφ. Διερωτώ με, σας ερωτώ, αν θα είσαστε γενική διευθύντρια της Όλαφ, τι θα κάνατε διαχειριστικά σε σχέση με την Όλαφ, τι θα κάνατε σε σχέση με τις 100 πρώτες ημέρες ως γενική διευθύντρια, ποια θα ήταν οι πρώτες σας, οι πρώτες σας, ποιες θα ήταν οι πρώτες σας προτεραιότητες. Ευχαριστώ οι πρώτε 100 μέρες. Εδώ ε, είναι σαν να μιλάμε για μήνα του μέλητο. Ε. Είναι η περίοδος που προσπαθεί κανείς ε, να εξοικειωθεί με το προσωπικό, με τους διευθυντές, αλλά και να δημιουργήσει σχέσεις με τους υπεύθυνους. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Διάβασα τις αιτήσει εκθέσεις, τις επικρίσεις ε, κατά της αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα ξεκινήσω ακούγοντας το τι έχουν να μου πούν. Θα προσπαθήσω να μάθω εάν το προσωπικό και η ηγεσία συμφωνεί με την άποψη που έχει το Κοινοβούλιο και η Εποπτική Επιτροπή για την ΟΛΑΒ. Γιατί νομίζω ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς όταν πρέπει να κάνει αλλαγές. Θα πρέπει να δούμε αν καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας. Δεν μπορεί κανείς ε, να δώσει εντολή για μια αλλαγή. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει κατανοητή. Τις πρώτες 100 μέρες λοιπόν θα ακούσω πολύ και μετά θα δράσω. Ευχαριστώ. Κύριε Ζόντεργκερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι τα προσόντα σας στον τομέα των φορολογικό είναι ιδιαίτερα ε, και πολύ καλά. Το επιχείρημά σας ε, για άλλες ε, εξεταστικές δραστηριότητες αφορά το επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας. Αναφερθήκατε στην διεθνή συνεργασία. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω για, το, για ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, γίνεται λόγος σε αυτό το πλαίσιο. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την ε, γραπτή σας δήλωση σε ένα θέμα. Εκεί αναφέρεστε και λέτε ότι επιθυμείτε η Όλαφ να γίνει γνωστή ως όργανο για την διαφάνεια με την οποία θα εργάζεται. Στα αγγλικά αναφέρεται θέλω για την διαφάνεια να γίνει γνωστή από πλευρά ιστεροφημία τη η Όλαφ. Αυτό σε τι αναφέρεται, στο παρελθόν ή στο μέλλον. Είναι μια ε, επίκριση όσον αφορά το καθεστώ διαφάνεια ε, της Όλαφ. Και τότε τι έχετε υπόψη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Α, δύο ερωτήσεις μου κάνατε. Η πρώτη αφορούσε τις ε, περιπτώσεις. Εγώ συνεργά, στον τομέα, στην εφορία για 20 χρόνια. Κάθε περίπτωση που καταλήγει στο τραπέζι μου μπορεί να ξεκινάει από τους φόρους, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο μέσα. Καταλαβαίνω ότι γνωρίζετε την δεκαετία του 20 και του 30, τότε που καταδικάστηκε οι καπώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν υποψίες ε, για διάπραξη φόνων, αλλά αυτό που τον οδήγησε στη φυλακή ήταν η φοροδιαφυγή. Αυτή είναι και η δική μου εμπειρία. Εργάστηκα, με απασχόλησαν πολλές περιπτώσεις που αφορούσαν και το οργανωμένο έγκλημα. Σε κάθε περίπτωση ενέχοντο, ναρκωτικά, βία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς στην καταδίκη μιας ομάδας, μιας συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος. Ε, ε, εκείνο που ελπίζουμε είναι να το συλλάβουμε ε, σε επίπεδο φορολογικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι αναγκαία για να κερδίσει κανείς το σεβασμό αυτών που βρισκόνται εκτός της οργάνωσης. Αν κάνει κανείς σωστά τη δουλειά του μπορεί να μην αρέσει στους άλλους. Εάν υπάρχει όμως διαφάνεια, αν είναι ξεκάθαρο το τι κάνεις και το πώς το κάνεις, τότε πιστεύω ότι ακόμα και μία οργάνωση που κάνει έρευνες όπως η όλα μπορεί να κατακτήσει το σεβασμό. Θα πρέπει όμως να υπάρχει διαφάνεια για να μπορεί κανείς να αξίζει αυτό το σεβασμό. Μάκοβεϊ. Ευχαριστώ. Έχετε ένα παρελθόν επιτυχούς διαχείρισης ε, περιπτώσεων απάτης και πραγματικά Εκτιμώ την απόφασή σας να υποβάλλετε υποψηφιότητα. Η πρώτη μου ερώτηση, η διαφθορά δεν είναι ένα θέμα που εντάσσεται στην εντολή της Όλαφ. Ξέρουμε όμως ότι η διαφθορά και η απάτη συνδέονται άρρηκτα μεταξύ του. Έχετε κάποιο πρόγραμμα, έχετε σκοπό να βρείτε αυτή τη σχέση μεταξύ τους και αυτό να μεθερμινευτεί σε περισσότερη δράση για την Όλαφ. Ποια είναι η άποψή σας για τη σχέση αυτή μεταξύ απάτης και διαφθοράς. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας της Όλαφ. Το ξέρουμε, το συζητήσαμε. Το πρώτο αφορά την έκταση των ερευνών. Τι θα κάνετε για να μειώσετε το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή μιας έρευνας. Πιστεύετε ότι μια λύση είναι να καθορίζονται προτεραιότητες και αν όντως το πιστεύετε με τι κριτήρια θα γίνει αυτός ο καθορισμός των προτεραιοτήτων. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τη διαφθορά. Δεν είναι συγκεκριμένο μέρος ε, της εντολής της Όλαφ. Πιστεύω ότι η Όλαφ θα ασχοληθεί πολύ με τα θέματα απάτης. Πιστεύω ότι ότι είναι ευθύνη της Όλαφ να προτείνει αλλαγές. Θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να εξετάσουμε την, ε, την εμπειρία που έχει η Όλαφ σε αυτό το τομέα για να διαπιστώσω εάν είναι καλή απόφαση την Όλαφ να προτείνει μια λύση στο νομικό ε, μια αλλαγή στο νομικό πλαίσιο. Τη δεύτερη ερώτηση αφορούσε το, τη διάρκεια των ε, ερευνών. Έχω σκοπό να θέσω προτεραιότητες. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, ναι, θα έλεγα ότι έχω. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που θα πρέπει, που μένουν ακόμα να εξεταστούν. Ο, η μέση διάρκεια μιας έρευνας ξεπερνάει τα δύο χρόνια. Κατά την άποψή μου αυτός ο μέσος όρος είναι απαράδεκτος, εντελώς απαράδεκτος και μόλον ότι η βεστιάζει την προσοχή της στις δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει μια συρρήκνωση του ε, χρόνου. Διαφορετικά δεν έχει κανείς να, τα κάνει, ε, να κάνει τα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να κάνει πολλά πράγματα παράλληλα. Το ένα θα ήταν να βρει δέκα ε, έρευνες και να τις χαρτογραφήσει και να προσπαθήσει να βρει τι είναι εκείνο που παρατείνει τα πράγματα. Ε, να εξετάσουμε αν υπάρχουν, αν έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα εργαλεία, πώς χρησιμοποιούμε την ανάλυση των κινδύνων, την πληροφόρηση, πώς ξεκινάμε τη δουλειά μας. Ξέρω ότι υπάρχει ένα εγχειρίδιο για όλα αυτά, αλλά εφαρμόζεται Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα με διάφορες δράσεις ε, για να μειωθεί η διάρκεια των ερευνών. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, κυρία Γιάλα Σέντερ. Κυρία ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, ε, κυρία Γκέλεμπραντ. Εσείς παρουσιάζεστε ως μια εξαιρετική διαχειρίστρια και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτό το είδος ε, χαρακτήρα χρειαζόμαστε. Όμως η Όλαφ είναι ένα μέσο που αντιμετωπίζει μια πρόκληση διαχειριστική και ποιοτική και ποσοτική για αυτή την πτυχή την ποιοτική θα ήθελα να ξέρω ποιο, ε, ποια άτομα ήταν εκείνα τα οποία εσείς είχατε ως ευθύνη στην ε, διαχειριστική σας δραστηριότητα ποσοτικά και ποιοτικά θα ήθελα να μας σχολιάσετε κάτι. Μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει αυτή η προσπάθεια, μια και οι ομάδες ε, είναι πολύ διαφορετικές και έχουν μεγάλο πολυσχηδές εύρος δραστηριοτήτων και θα ήθελα να ξέρω σε σχέση με τις προθεσμίες τι θα γίνει. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το, η, μέση, η μέση περίοδος ε, για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων από το γραφείο σας. Θέλουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η διάρκεια των ε, ερευνών ε, και πώς το βλέπετε εσείς. Και το most noticeable personal θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι αυτό που είπατε, θα ήθελα να αντιμετωπίσω την απάτη με ένα θαυμαστικό με που ακολουθεί. Με ενθουσιασμό και ζήλο ε, αντιμετωπίζεται αυτή την ε, προοπτική. Όμως η Όλαφ είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να καταστρέψει την ιστεροφημία ατόμων ε, και θα ήθελα να ξέρω με ποιο, ποιο είδους δεοντολογικό κώδικα θα δράσετε για να αποφευθούν τέτοιου είδους, ας το έτσι, ολιστήματα. Ευχαριστώ. Uh, και τέσσερα ερωτήσεις. Ας δω αν τις θυμάμαι όλες τώρα. Σχετικά με την ποιότητα και το μέγεθος των ομάδων. Αυτή τη στιγμή ε, είμαι πριν μια οργάνωσης με 2.000 άτομα, τα οποία χωρίζονται σε ομάδες, σε 12 διαφορετικά γραφεία και τα γραφεία επίσης υποδιαιρούνται σε τμήματα 20 ατόμων το καθένα και οι ομάδες έχουν μεταξύ δύο και 4 ατόμων. Λοιπόν, για την καθημερινή μου δραστηριότητα. Εγώ έχω την διαχειριστική ομάδα, 8 άτομα. Όταν όμως παρακολουθώ, κάνω το follow-up και βλέπω τα αποτελέσματα, ε, συναντώ τους διευθυντές μου και τότε μαζευόμασταν 100. Κάθε δύο μήνες συγκεντρωνόμαστε όλοι οι διευθυντές συγκεντρώνονται οι διευθυντέ των 12 γραφείων μαζί με τη διαχειριστική μου ομάδα, την ομάδα διοίκηση, δύο φορέ το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ασκώ τη διοίκηση μέσω των άλλων. Τώρα για το πολιτισμικό περιβάλλον και την ποικιλότητα μέσα στην, και τη διαφοροποίηση μέσα στην ε, ομάδα. Σήμερα στην οργάνωσή μου έχω μεταξύ περίπου 20%-30% ε, των ατόμων που εργάζονται σε εμάς προέρχονται από άλλες χώρες εκτός της Σουηδίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργαζόμαστε με άτομα από άλλες χώρες. Το πλεονέκτημα είναι ότι όταν γίνεται ένας έλεγχος σε μια επιχείρηση δεν ακούω πια παράπονα ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, ότι δεν καταλαβαίνουν την κουλτούρα, επειδή συχνά ε, γίνονται έλεγχοι στη γλώσσα του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Δεν είναι εύκολο, πράγματι δεν είναι εύκολο να δικεί κανείς μια οργάνωση πολυπολιτισμική. Πρέπει κανείς να είναι υπομονετικός. Έχω δημιουργήσει ένα πρόγραμμα δίκησης για τους διευθυντές με βάση μια μελέτη της Ολλανδίας, έναν καθηγητή ονόματι Hofstadter, που έχει ως αντικείμενο να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί τις διάφορες κουλτούρες και γλώσσες που έχουμε στην οργάνωσή μας. Αυτό έχει στεφθεί με επιτυχία. Αυτό όμως γίνεται με τα χρόνια, ε, δεν γίνεται νυχθημερών. Κατόπιν ένα ερώτημα σχετικά με τις προθεσμίες. Σήμερα και εμεί έχουμε, στη δική μου την οργάνωση, έχουμε να κάνουμε περίπλοκε περιπτώσει, όπω και η Όλαφ. Οι περίπλοκε περιπτώσει είναι εκείνε τι οποίε αντιμετωπίζουμε και εξετάζουμε με την εισαγγελία και την αστυνομία. Εμεί έχουμε προθεσμία 10 μηνών. Το 80% των περιπτώσεων θα πρέπει να έχουν επιληθεί μέσα σε 10 μήνε. Διαφορετικά, θα πρέπει προσωπικά να λογοδοτήσουν σε μένα και να μου εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν λύθηκε το θέμα. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Εδώ και πέντε χρόνια έχουμε αυτό το σύστημα και επιτελείται πρόοδο κάθε χρόνο. Αλλά και πάλι θα πρέπει να είσαστε υπομονετικοί, να επιμένετε, διαφορετικά δεν θα υπάρχει συνεχής πρόοδο. Νομίζω ότι μου τέθηκε ένα ερώτημα που είχε σχέση με τον κώδικα διοντολογίας στην οργάνωση που διευθύνω. Είχαμε πριν από 10 χρόνια αποφασίσει για τη διοντολογία που, θα, που θέλουμε ε, να εφαρμόσουμε για την καθημερινή μας δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να εξηγήσετε στα άτομα. Πρέπει να είναι κάτι που αισθάνεστε για να το μεταφέρετε. Πάλι, αυτό δεν είναι κάτι το εύκολο. αισθάνεται κανείς μεγάλη ικανοποίηση όταν ε, καρποφορήσουν οι προσπάθειές σου. Αλλά χρειάστηκαν τρία-τέσσερα χρόνια πρωτού πω πραγματικά ότι το προσωπικό μου είχε καταλάβει ε, τι σήμαινε ο δικός μας κώδικας δεντολογίας. Ε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι δυνατόν. Sorry, Δεν έκανα λόγο για τον εσωτερικό κώδικα εργασιών, αλλά για τον δεοντολογικό κώδικα σε σχέση με τα άτομα και τις επιχειρήσεις που αφορώνται από αυτές τις εξεταστικές δραστηριότητες. Συγχωρείτε, δεν το κατάλαβα καλά, με συγχωρείτε. Όταν κανεί δηλαδή ενέργεια έρευνα διοικητικού επίπεδου ή αστυνομικού επίπεδου, όταν συνεργάζεστε με αστυνόμο ή εισαγγελέα, πρέπει να φροντίσετε ότι συνεργάζονται σωστά αυτοί οι τρεις. Και φυσικά τα άτομα έχουν δικαιώματα τα οποία εξετάζετε, διερευνάτε και πρέπει λοιπόν να φροντίζετε οι έρευνες να διενεργούνται με τρόπο που να σας επιτρέπουν να εφαρμόζετε τον κώδικα ηθικής δεντολογίας και τη νομική διάρθρωση που απαιτείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Thank Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Γκέλεμπραντα, πολλά υπόθηκαν σχετικά με την ισορροπία μεταξύ του ερευνητικού και του δικαστικού ρόλου της Όλαβα. Τίποτα όμως δεν υπόθηκε για το θέμα της κράτησης. όχι. Διερεύνηση. Πιστεύετε ότι καμία ανακριτική εργασία δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει αυτή η διερεύνηση. Και αυτό είναι κάτι που μέχρι τώρα έχει αμελήσει η Όλαφα. Και αν συμφωνείτε με αυτό, πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο τομέας. Well, of course, you have to detect the fraud and find it first, otherwise you can't <laughs> investigate it. So you're absolutely right. Thank you for asking me that. Πρέπει να ανοιχνεύσετε πρωτού κάνετε οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το 50% των ερευνών uh, της Όλαφ σήμερα ξεκινάν με τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Πιστεύω ότι η Όλαφ θα πρέπει να προβλέπει τις καταστάσεις κατά κάποιο τρόπο διότι θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνων και να σκεφτεί πού κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να εκδηλωθεί απάτη. Πρέπει να προβλέψετε το κακό, διαφορετικά δεν μπορείτε να το ανοιχνεύσετε. Και παρόλο ότι όλα είναι πολύ καλή οργάνωση, διότι έχει ε, αυτή την πολυ, πολιτισμική και πολυτομιακή διάρθρωση, ομάδες που είναι αρμόδιες για πολλούς τομείς, έχουν εισαγγελίες, έχουν άτομα με νομική και οικονομική εκπαίδευση. Για να ανοιχνεύσετε την απάτη, να τη βρείτε την απάτη, πρέπει να έχετε τέτοια κατάρτιση. Αλλά επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε και όλα τα σύγχρονα μέσα για να μπορέσετε να διαπιστώσετε, να βρείτε ε, την απάτη και να την καταπομελεμήσετε με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία μου, κυρία Γκέλεμπραντ, τελειώσαμε για σήμερα με τις ακροάσεις. Ευχαριστώ. Θα ξαναρχίσουμε αύριο το πρωί στις